Okay, colleagues, uh, we'll begin the meeting. So, colleagues, we're going to begin. Παρακαλώ, Καλό σας απόγευμα. Αρχίζουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε τις εξής αλλαγές. Ένα νέο σημείο 3α, αναπομπή στην Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 69.3 σε σχέση με τους καταλόγους ε, πολιτών τρίτων χωρών που θα πρέπει να διαθέτουν θεωρήσεις ως προς τα εξωτερικά σύνορα με βάση την απόσυση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα γίνει από τις 7 και 10 μέχρι τις 7 και 20. 7 και 20 αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στην ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Ανακοινώσει του Προέδρου έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από δανέζικα, κροατικά, μαλτέζικα και κελτικά. Δυνάμει του άρθρου 205 ως προς τους συντονιστές έχουμε το feedback των συντονιστών της 27ης Φεβρουαρίου. Θα το δείτε αυτό στις ε, ανακοινώσεις σας. Ο κύριος Φρανς θα αντικαταστήσει τον κύριο Άλμπρεχτ στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το ΕΝΙΣΑ, ε, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και η Άννα Μιράντα έχει διοριστεί συγγήτρια για το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020. Εγκρίνεται, ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει στις 7 και 20 να έχετε τις κάρτες σας παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η αναπομπή στην Επιτροπή σε σχέση με την προσωρινή επανεισαγωγή, ε, μάλλον επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά ε, σύνορα. Η κυρία Τάνια Φαγιόν δεν είναι ε, παρούσα. Η κυρία Σίπελ, Σίπελ θα μας κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας διαβάσω ορισμένες ανακοινώσεις της Τάνια Φαγιών. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 29 Νοεμβρίου 2018 η Ολομέλεια ενέκρινε τρόπο σε σχέση με τον κώδικα του χώρου του Σέγγεν σε σχέση με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και ανέπεμψε το θέμα στη Λίμπε. Είχαμε δύο τριμερεί στις 12 ε, Δεκεμβρίου και στις 13 Ιανουαρίου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ρουμανικής Προεδρίας πήγαν πολύ καλά. Παρά όμως το γεγονός ότι θέλαμε μέχρι το τέλος της θητείας να εγκρίνουμε τον κανονισμό, είχαμε μία αναπέμπουσα ε, μειοψηφία, αναστέλουσα με συγχωρείτε μειοψηφία και γι' αυτό στις 8 ε, Φεβρουαρίου η κυρία Λουμινίτσα Ορομπέσκου, η πρέσβης, ε, ανέφερε στην ε, Τάνια Φαγιόν ότι δεν θα μπορούσε να περάσει η απόφαση της ε, Κόρεπερ του 2018 και ανεστάλησαν οι διαπραγματεύση. Η Τάνια Φαγιόν θεωρεί ότι χρειάζεται αυτή η προσωρινή επαναφορά. Έχουμε έξι κράτη-μέλη του χώρου του Σέγγεν που ε, διατηρούν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και αυτό που είναι πιο ανησυχητικό είναι ότι έξι αυτές χώρες ε, έχουν παρατεταμένους ελέγχους παρά την διετή περίοδο που έχει ορίσει η Επιτροπή και η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέτρα εναντίον τους. Παρόλα αυτά, έχω έχουμε μεγάλη μείωση νέων ε, προσελεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο ε, προς το συμφέρον ευρωπαϊκών ε, κυβερνήσεων, κάτι το οποίο κατακρίνει η συνάδελφος Τάνια. Παρά τις προθέσεις μας δεν μπορέσαμε να άρουμε το αδιέξοδο. Οι ομάδες μας καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να γίνει κάποια πρόοδος και η Τάνια τους ευχαριστεί ιδιαίτερα. Τέλος, λάβοντας υπόψη τις θέσεις των σκιωδών, η Τάνια έφτασε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη επιλογή για το Κοινοβούλιο θα ήταν να κλείσει η πρώτη ανάγνωση με βάση την εντολή της Ολομελίας της 29 Νοεμβρίου 2018. Γι' αυτό το αίτημα της Τάνια προς τη Λίμπε και τον Κλοντ είναι το θέμα να τεθεί στην ε, ε, ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας έτσι ώστε να έχουμε μια ενιαία διαδικασία και να κλείσει και η πρώτη ανάγνωση. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Μπίργκιτ. Συνάδελφοι, έλαβα ένα mail στη, την 5η Μαρτίου και ζητήθηκε από τη ΛΥΜΠΕ, από τους συντονιστές και τα μέλη να εισαχθεί το θέμα αυτό στην Ολομέλεια για μία και μοναδική ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα ενημερώσω τον Πρόεδρο, δηλαδή ενία πλειοψηφία στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης και των τροπολογιών που ενεκρίθησαν τον Νοέμβριο. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις τότε θα το υποβάλουμε στους συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλα θέματα. Όχι. Ευχαριστούμε Birgit για τις θέσεις της κυρίας Φαγιών που μας τις κοινοποίησες. Ωραία. Τώρα έχουμε το 3α που είναι ο κατάλογος τρι, τρίτων ε, χωρών και πολιτών που πρέπει να ε, κατέχουν, να έχουν μάλλον ε, θεωρήσεις. Συνάδελφε, συνάδελφοι, από τότε που ψηφίσαμε στις 29 Ιανουαρίου, ε, ομόφωνα με 53 τρεις ψήφους εγκρίναμε το πλαίσιο και είχαμε τρεις ε, 3, 6 και 27 Ιανουαρίου. Ένας πέμπτος θα γίνει στις 12 Μαρτίου, αύριο δηλαδή, μετά τις 6, 12, 20 και 27. Ξέρω ότι θέλετε να συζητηθεί το θέμα, μπορώ να σας ε, πω πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ένας πέμπτος ε, τριμερής θα λάβει χώρα αύριο. Έχουν ε, συναντηθεί οι τριμερείς. Πόσο έχουμε για αυτό το θέμα? Δέκα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά επειδή πολλοί θέλουν να λάβουν το λόγο, θα το παρατείνουμε για να μιλήσουν όλοι, εάν θέλετε να λάβετε το λόγο. Ο πέμπτος τριμερής θα γίνει αύριο. Για να σας επεξηγήσω, στην τελευταία συνεδρίαση σας είπαμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα άλλα ζητήματα. Καθίσταται σαφές ότι το θέμα αυτό είναι περίπλοκο. Το η υποσημείωση δείχνει ότι μετά από τέσσερις τριμερείς και πέντε διαφορετικές διατυπώσεις προς το Συμβούλιο δεν υπήρχε νομική απέτηση για να μπει αυτή η υποσημείωση για ένα φάκελο που έχει σχέση με τις θεωρήσεις. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Όμως ε, ανέκυψε ένα πολιτικό ζήτημα όπου μία χώρα έθεσε υποσημείωση και άλλαξε τη θέση του Συμβουλίου και κράτησε τη θέση του. Μετά από τέσσερις τριμερείς και πολλές προσπάθειες να φτάσουμε σε μια εναλλακτική διατύπωση. Διατύπωση η οποία χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατα άλλα ζητήματα για το Brexit όπου αναφέρεται το Γιβραλτάρ παρά αυτά τα προηγούμενα καταλαβαίνουμε ότι έγιναν πολύ περιορισμένες συζητήσεις στο Συμβούλιο. Όμως ε, μπορώ να σας πω ότι έγιναν ορισμένες συζητήσεις στο Συμβούλιο και αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στον πέμπτο τριμερή διάλογο. Δεύτερον, με τον πέμπτο τριμερή τα τρία θεσμικά όργανα και εγώ ως και οι που θα να τους ευχαριστήσω για την υπομονή τους γιατί φτάσαμε σε συγκεκριμένα πολιτικά συμπεράσματα ε, γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να εγκριθεί η διαδικασία θεωρήσεων και μετά τη συνάντηση των σκιωδών αυτό ακριβώς άκουσα, άρα έχουμε ένα πέμπτο τριμερή και ελπίζω ότι στο πέμπτο τριμερή διάλογο θα έχουμε άρση του αδιεξόδου μετά τον πέμπτο τριμερή και αυτό το συζήτησα με του σκιώδεις, Καταλαβαίνετε ότι τελειώνει και ο χρόνος μας για τις θεωρήσεις. Άρα τα ουσιώδη ζητήματα δεν έχουν αλλάξει. Η εισδοχή του υποσημειώματος δεν έχει αλλάξει. Οι Ισπανοί έχουν σαφή θέση επί του θέματος και το θέμα αφορά και τον θεσμικό εισηγητή. 53 ψήφους υπέρ, κανείς κατά. Πέντε προσπάθειες έγιναν για την εναλλακτική εντύπωση αναφέροντας το Γιβραλτάρ. Αυτό έγινε ως προς το Brexit. Αύριο ελπίζω να τα καταφέρουμε και η Επιτροπή προτείνει, θα προτείνει και κάτι άλλο για αύριο. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά ελπίζω να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει. Γιατί η θέση του Συμβουλίου είναι πολιτικής υφής καθαρά. Δηλαδή είδα τη μία διατύπωση μόνο. Ωραία. Αρχίζουμε τώρα το διάλογο. Έχω. Λόπες Αγγιλάρ. Mr. Diaz and Maita. So we start with uh, Mr. Lopez Aguilar. If everyone can stick to two minutes. Αν θέλετε να μείνουμε στα δύο λεπτά, συνεχίζει ο Πρόεδρος, παρακαλώ ο κύριος ε, Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Κλόντ. Πολύ σύντομα. Εκτιμώ το θεσμικό σου ρόλο ως προ, πρόεδρος και ως συντονιστής όλης αυτής της προσπάθειας της δουλειάς. Εκτιμώ την προσπάθεια που κάνεις, επαναλαμβάνω. Έχουμε όμως κάνει τρεις τριμερείς διαλόγους σε ένα φάκελο που δεν θα έπρεπε καθόλου να είναι προβληματικός, εκτός από το σημείο στο οποίο αναφέρθηκες που δεν είναι περιθωριακό συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν να κινούνται οι πολίτε χωρί θεωρήσει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα, γιατί έχουμε μπλοκαριστεί τρεις τριμερείς διαλόγους τώρα και γιατί περιμένουμε να ξεμπλοκαριστούμε στον πέμπτο ίσως. Διότι υπάρχει μια θέση που ειναι το προβλημα γιατι εχουμε μπλοκαριστει τρει τριμερει διαλόγου τωρα και γιατι περιμενουμε ομόφωνα 27. Τα 27 κράτη-μέλη και που υποστηρίζεται και στην ε, δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπής ότι δηλαδή καμία εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου δεν θα μπορεί να γίνει που να επηρεάσει το Γιβραλτάρ. Εάν δεν προχωρήσουμε αύριο, η μόνη λύση θα είναι να πούμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα επίλυσης διότι η θέση του συμβολίου δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου. Μιλούμε για τη δυνατότητα απολύτως εντός των κανόνων να διευκολυνθεί το όνομα του εισηγητού. Δεν υπάρχει συνθήκη προϋπόθεση να είναι υπήκος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά είχε λεχθεί με σαφήνεια ότι δεν θα πρέπει το άλλο πρόσωπο να είναι από την άλλη ενδιαφερόμενη χώρα που είναι το βασίλειο της Ισπανίας. Εντάξει. Αλλά πρέπει οι συντονιστές να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτό. Διότι αλλιώς μία οδός που φαίνεται να οδηγεί σε μια επίλυση δεν θα ολοκληρωθεί. Δεν θα καρποφορήσει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιέζεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης της Άλντε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς συναδέλφους που όσες εισηγητές υπερασπίστηκαν θαραλέα τη θέση αυτής εδώ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Αλλά είδαμε το Συμβούλιο να είναι ενωμένο και το Κοινοβούλιο όχι. Οι συνάδελφοι προσπάθησαν θεραλέα μέχρι το τέλος, είτε για τον μηχανισμό για τις θεωρήσεις, είτε για άλλα θέματα και επέτυχαν κάποιες συμβαστικές λύσεις. Και τώρα μας λένε ότι θα πρέπει να δεχθούμε τη θέση του Συμβουλίου ως έχει. Δεν το καταλαβαίνω. Πέντε συμβαστικές προτάσεις αποστήλαμε στο Συμβούλιο και στην αρχική μας θέση 53-02 δεν υπήρχε καμία αναφορά στο Γιβραλτάρ. Στις συμβασικές μας προτάσεις προχωρήσαμε, κάναμε πολλά βήματα προς την πλευρά του Συμβουλίου ώστε να υπάρξει ρητή αναφορά στο Γιβραλτάρ το οποίο ήταν ε, ξεκάθαρη υποχώρηση προς το μέρος του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο όμως εξακολουθεί να λέει όχι, όχι, όχι. Και νομίζω ότι η Προεδρία δεν το συζητεί σοβαρά αυτό στο Συμβουλίο. Δεν συζητεί σοβαρά την πρότασή μα, τι προτάσει μα, οι οποίε προσπαθούν να προσαγγίσουν το Συμβουλίο. Εγώ βλέπω ότι αυτό είναι προσβλητικό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέσσερις τριμερεί διάλογοι, το Συμβούλιο δεν συζητά, δεν μας θεωρεί σοβαρού συνομιλητέ. αυτό είναι προσβολή. Διάθετη μέρο, παρακαλώ. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η θέση μου είναι γνωστή. Δεν θα επαναλάβω. Υπήρξε σαφής νομίζω στην ε, προηγούμενη συζήτηση και σε σχέση με νέα επιχειρήματα, Πρόεδρε, εσείς λάβατε 53 ψήφους εντολής, μεταξύ των οποίων τη δική μου, Αλλά όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, η νομοθετική διαδικασία εξαρτάται και από τα δύο θεσμικά όργανα. Και το Συμβούλιο ομοφόνος, 27 27-1 1, ρητή συμφωνία της Ισπανίας λέγει έχουμε ένα αμφίσιμο ζήτημα, ένα αντιφατικό ζήτημα και λέει το Γιβρατάρ είναι απικία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη σημεία αυτό και μετά δεν νομιμοποιείται η θέση σας. Γιατί δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τη θέση σας ως εισηγητού από τη θέση σας ως Βρετανού υπηκόου. Και επομένως έχουμε σύγκρουση αρμοδιότητος. Και αυτό αναφέρθηκε και στους προέδρους και από διάφορα άλλα μέλη του σώματος. Και υπάρχει και, ε, για να μην αναφερθώ σε ένα <laughs> θεμελιωδέστατο ζήτημα που είναι η ηθική. Υπάρχει ένα πρόβλημα και τέτοια φύσεως. Πρέπει να δώσετε τη θέση σας σε κάποιον που να μην είναι ούτε Βρετανός ούτε Ισπανός, ώστε να μην έχει αυτή τη σύγκρουση αρμοδιότητα, Πρόεδρε. Τίποτε άλλο. Μάλιστα, κύριε Ντία. Μάιτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας άκουσα όλους σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε και νομίζω ότι ε, τίθενται ε, δύο ζητήματα. Ουσίες αλλά και διαδικασίες Φαίνεται, δείχνει να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση στην οποία αντιπαρατίθενται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αλλά αγαπητέ Πίτερ, δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Είναι αλλά όχι ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι το Συμβούλιο έχει μία θέση που υποστηρίζεται πολιτικά ε, επαρκέστατα και τοποθετείται σχετικά με το συμφέρον του να αναγνωριστεί, μάλλον την αναγκαιότητα του να αναγνωριστεί η θέση αυτή που εκφράζεται η πολιτική επίσημα πρέπει να υπερασπίσει να κανείς ε, το, ε, ένα, ένα, ένα συμφέρον, μια θέση που έχει μια πολιτική και μια νομική διάσταση και επομένως με όλο το σεβασμό προς τους συναδέλφους. Εάν το Συμβούλιο υποβάλει μια πρόταση που είναι λογική, διότι πολιτικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα κράτος μέλος και για τη σχέση του με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή, διότι αυτό που προτείνει το Συμβούλιο είναι λογικό. Ε, η κυρία Σίπολα και μετά πρέπει να πάμε σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να συμμετάσχω στη συζήτηση, αλλά πρέπει να πω πως έχω μπερδευτεί κάπως διότι ήδη στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής μας ακούσαμε ότι οι συντονιστές, όλοι ψήφισαν ώστε ο πρόεδρος να αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν αφορούν συζήτηση για το νομικό καθεστώς του Γιβραλτάρ. Θα συζητηθεί η συνέχεια μετά το Brexit και αυτό που προσπαθούμε είναι να διασφαλίσουμε ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Ε, και τώρα ακούω για σύγκρουση συμφερόντων, αρμοδιοτήτων, όμως ε, οι περισσότεροι από όσους το είπαν είναι Ισπανοί. Αυτό δεν καθιστά από μόνο του σύγκρουση συμφερόντων. Και δεν νομίζω πως είναι δίκαιη λοιπόν αυτή η συζήτηση. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ούτε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε διατύπωση για περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ. Αυτή η διατύπωση ήταν του Συμβουλίου. Τώρα για ποιους λόγους δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Επιτροπής, ο εισηγητής και οι σκιώδεις έχουν κάνει μέχρι τώρα εξαιρετική δουλειά και προσπάθησαν να κρατήσουν τη θέση της Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου και να την αντιτάξουν απέναντι σε εκείνη του Συμβουλίου. Θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία αύριο να συνεχίσουν. Ο πρόεδρος ήδη μας είπε πως από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδεχομένως υπάρξει μια διάθεση συμβιβασμού. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας πάνω σε αυτά που ψηφίσαμε ως Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τοποθετηθεί, όμως σας υπενθυμίζω πως πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρέπει να ψηφίσουμε, γι' αυτό ας μην μπερδέψουμε τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους και σας ευχαριστώ πολύ που κρατήσατε τα πνεύματα ήρεμα από την τελευταία φορά. Επίσης, σε ό,τι φορά την απάντηση σε αυτά που ο κύριος Δίας μέρα, να πω πως έχω απόλυτη επίγνωση του πόσο δύσκολη πολιτικά είναι αυτή η κατάσταση. Ο στόχος, ο δικός μου και των σκιωδών εισηγητών, είναι να προσπαθήσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο το συντομότερο. Να το κάνουμε αυτό ε, με την ιδιότητα του θεσμικού εισηγητή ανεξαρτήτως εθνικότητας. Η δουλειά μας λοιπόν, η δουλειά μου είναι να υπερασπιστούμε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαφορά το Γιβραλτάρ και να σας πω εδώ ότι η Προεδρία δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Το Συμβούλιο έχει κάνει επίσης ελάχιστα πράγματα για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε έναν συμβιβασμό. Δεν, δεν υπήρξε καμία τέτοια προσπάθεια από το Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν στην ουσία προχωρούσαμε χωρίς να είμαστε σίγουροι για τίποτα. προχωρούσαμε χωρίς καμία ένδειξη προθέσεων. Είχαμε προτείνει πέντε λύσεις για το Γιβραλτάρ. Και όλες αυτές οι προτάσεις θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Συμβούλιο και όχι από μένα. Η δική μου γραμμή είναι ξεκάθαρη λοιπόν. Αύριο, όπως είπαν και οι Ισπανοί συνάδελφοι, εξαιτία των πολιτικών ζητημάτων που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε πλέον ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιληθεί το ζήτημα, να βγούμε από το αδιέξοδο. Και να ευχαριστήσω εδώ τους ε, σκιώδει ηγητές που μπήκαν και αυτοί στην πρώτη γραμμή και σκάγια για αυτήν την προσέγγιση που ήταν πάρα πολύ ενωμένη, έτσι ώστε να δοθεί μια λύση στον πέμπτο τριμερή διάλογο. Κάποιο από εσά είπε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι εύκολο και να το ολοκληρώσουμε πολύ γρήγορα. Ακριβώς γι' αυτό ανατέθηκε σε μένα θεσμικά, γιατί αναμενόταν να το είχαμε ολοκληρώσει μέσα σε τρεις μέρες. Αλλά το Συμβούλιο είναι εκείνο που δυσκόλεψε τα πράγματα και όχι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν να σας ευχαριστήσω ξανά για την συνεισφορά σας και για τις ε, τοποθετήσεις σας. Θα τις λάβω υπόψη στον ε, επόμενο τριμερή διάλογο. Αλλά τώρα νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες. If everyone is ready. Αν είστε όλοι έτοιμοι, μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. εισηγητής είναι ο κύριο Ντεπρέ. Θα θέλατε να πάρετε το λόγο πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τους σκιώδεις για την ποιότητα Τη συνεισφορά και την καλή ανταλλαγή απόψεων παρά τις διαστάσεις απόψεων. Ελπίζω η πλειοψηφία να συμφωνήσει γιατί βασιζόμαστε σε τέσσερα στοιχεία. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν κυρίαρχα για να δώσουν, να χορηγήσουν ή όχι ταυτότητες. Δεύτερον, ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να ταχθεί υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας με ένα ενιαίο πλαίσιο, format, που θα αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη με βιομετρικά στοιχεία που ε, επιτρέπουν την ε, αύξηση των προδιαγραφών ασφαλείας για να μην, ε, υπάρχει, να μην υπάρχουν σφετερισμοί. Δεν χρειάζονται εθνικές τράπεζες δεδομένων, αλλά θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Η θέση σε εφαρμογή θα αφορά την ισχύ των ε, ε, εγγράφων αυτών για να μην υπάρξει επιπρόσθετο κόστος για τα κράτη-μέλη και για τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεπρέ. Περνάμε στην ψηφοφορία λοιπόν, συνάδελφοι. Μία ψηφοφορία για το κείμενο που έχει συμφωνηθεί κατόπιν των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ, 20 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια, κύριε Ντεπρέ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την αναδιατύπωση σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιωματικών Συνδέσμων Μετανάστευση. Η συγγήτρια είναι η Σεσίλ Κέγκε. Θα θέλατε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κλώτα. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με μεγάλη ευθύνη, επαύξησαν το ρόλο ε, του γραφείου συνδέσμου. Έχουμε λοιπόν μια νέα ψηφίδα στην πολιτική χορήγηση ασύλου και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσσωμο ενέκρινε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ του Σκιώδης αλλά και τη Γραμματεία για τη σύνδρομή της. Ευχαριστούμε πολύ, Σεσίλ. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Άρχεται. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία τον εξουσιο... σε κανονισμό της Επιτροπής για τροποποίηση του παρατήματος 2 του κανονισμού 515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας του Μέσου Χρηματοδοτικής στήριξη στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια και έπειτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Ζίπελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ακούσω την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς την πρόταση, γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να τους ακούσουμε. Πολύ ωραία. Κύριε Ονίδη. Αν θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Ζήπελ, μπορείτε να προχωρήσετε πρωτού περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Με συγχωρείτε που καθυστερώ την ψηφοφορία σας. Να πω λοιπόν ότι αυτές οι κατεξουσιοδότηση πράξεις έχουν έναν στόχο, να τροποποιήσουν δηλαδή τις αντίστοιχες νομικές βάσεις έτσι ώστε να επιτρέψουν την κατάλληλη χρηματοδότηση του, ε, των κέντρων υποδοχής στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται έτσι ώστε να επιτρέψουμε στο πλαίσιο της ESTIA, να υπάρξει κατάλληλη στέγαση και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά και να ε, υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν τα κέντρα αυτά. Και λυπούμαστε πάρα πολύ για τη σύγχυση που έχει επέλθει σχετικά με αυτές ε, τις τροποποιημένες πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Η έννοια του, των ελεγχόμενων κέντρων έχει εισαχθεί στο κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους μας να χρησιμοποιήσουμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση για να χρηματοδοτήσουμε τα αποκαλούμενα κέντρα ελέγχου προτού εκείνα προτού μάλλον καθοριστεί η λειτουργία τους. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε αυτά τα κέντρα να είναι σαφώς ε, δημιουργημένα και να είναι σε ξεκάθαρη λειτουργία τους. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ε, ομαλή λειτουργία των κέντρων υποδοχής στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεσή μας να παρακάμψουμε την ε, αρμοδιότητά σας για να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης αυτών των κέντρων ελέγχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, Μπίργκιτ, θα ήθελες να απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε μεγάλη προσοχή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πάλι είμαι κάπως μπερδεμένη. Ίσως οι προθέσεις σας να μην είναι παράλογες, όμως ε, ο ορισμός κέντρα ελέγχου υπάρχει στην πρόταση. Με αυτή τη διατύπωση κανείς δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Επίσης αναφερθήκατε σε κέντρα υποδοχής, reception centers, αλλά αν ε, θέλετε να μιλήσετε για κέντρα υποδοχής, γιατί δεν τα λέτε έτσι, γιατί αναφέρεστε σε κέντρα ελέγχου. Αυτό μου φαίνεται κάτι καινούργιο που εισάγεται εδώ και ίσως οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση μπορεί να βοηθούν και να εξυπηρετούν στο σκοπό σας, όμως βλέπουμε ότι για μία ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ανακατέψει τα πράγματα έτσι ώστε να εφαρμόσει πράγματα και να υλοποιήσει τις δικές της προθέσεις με την διατύπωση κέντρα ελέγχου ο καθένας μπορεί να νομίζει ό,τι θέλει, να το τροποποιήσει κατά το δοκούν. Δεν είχαμε λοιπόν τον ε, κατάλληλο χρόνο για να ελέγξουμε ε, το περιεχόμενο και το τι σημαίνει αυτός ο ορισμός, κέντρα ελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι λίγο περίπου που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα για αυτήν την πράξη κατά εξουσιοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατόπιν όλων αυτών, της απάντησης της Επιτροπής και της ε, τοποθέτησης της ηχήτριας θα ψηφίσουμε δύο φορές. Ξεκινάμε με την πρώτη ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους υπέρ 8 κατά και καμία αποχή. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Άρχεται. Και πάλι ε, για το σημείο 7, με την κυρία Σίπελ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 44 ψήφους υπέρ 8 κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα, κυρία Ζήπελη. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε τώρα σε άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο, το σημείο 8. Και αγαπητοί συνάδελφοι, αν μείνετε πολύ ε, καλώς, αν φύγετε, να αποχωρήσετε ήσυχα, γιατί έχει έρθει η ώρα για την ακρόαση υποψήφια που έχει επιλεγεί για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Συνάδελφοι, παρακαλώ, αποχωρήστε ήσυχα αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μείνετε, αν μπορείτε, διότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνάδελφοι, να καλωσορίσω λοιπόν στην Επιτροπή μας την κυρία Νίνα Γκρεγόρη, την υποψήφια που έχει επιλεγεί. Παρακαλώ, αποχωρήστε ήσυχα. Την υποψήφια λοιπόν, κυρία Νίνα Γκρεγόρη, που έχει επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέση της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Η κυρία Γκρεγόρη θα κάνει μια δήλωση και θα απαντήσει σε ερωτήσεις ε, των μελών της Επιτροπής πριν τον διορισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού της ΕΑΣΟ. Κανονισμού 439 ε, του 2010. Επίσης, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων και των εισηγητών θα απαντήσει η κυρία Γκρεγόρη στις ερωτήσεις μας. Κατόπιν τούτου, οι συνάδελφοι θα διατυπώσουν τη, τη σύστασή τους για την υποψηφιότητα της κυρίας Γκρεγόρη και κατά την προετοιμασία αυτής της ακρόασης υποβάλαμε γραπτές ερωτήσεις στην κυρία Γκρεγόρη, λάβαμε τις απαντήσεις ε, της μπορείτε να βρείτε τόσο τις απαντήσεις όσο και το βιογραφικό της κυρίας Γκρεγόρη στον ιστότοπο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρεγόρη για να μας ε, κάνει την παρουσίασή της εντός 10 λεπτών και μετά θα περάσουμε στις τοποθετήσεις των εισηγητών και τις ερωτήσεις όλων των υπόλοιπων συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Γκρεγόρη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη της ΛΥΠΕ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον σας ως εκλεγμένη ε, υποψήφια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΖΟ. Βεβαίως, ε, ε, σας απάντησα και γραπτός, όπως είπε ο Πρόεδρος, θα ήθελα όμως να σας πω ποια είμαι, να σας κάνω μία εισαγωγή και να σας <clears throat> μιλήσω για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσω καθώς και το όραμα για, για τον οργανισμό αυτό. Προέρχομαι από τη Σλοβενία και έχω ο εργαστής στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου στο Υπουργείο Εσωτερικών τα 20 τελευταία χρόνια. Τα 10 <coughs> τελευταία χρόνια ήμουνα Γενική Διευθύντρια ε, στα πλαίσια του Εθνικού Οργανισμού Ασύλου. Μετά από 10 χρόνια διευθυντικής θέσης έδειξα την ηγετική μου θέση και την δυνατότητα αντιμετώπισης στρατηγικών ζητημάτων και διοικητικών καθώς ε, και δημοσιονομικών καθώς και θέματα ε, ανθρώπινων πόρων. Από το 1999 και εξής ασχολήθηκα με τη σλοβενική θέση από πλευράς ε, εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης και ήμουνα επικεφαλής της ομάδας ΚΙΦΑ που ασχολείται με θέματα ασύλου στα σύνορα. Ε, έχω, ε, ήμουνα υπεύθυνη μάλλον σε 10 επιτροπές και διοικητικά συμβούλια και έχω παραστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πολλές φορές. Άρα έχω μία σφαιρική πολιτική κατανόηση του θέματος. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης ε, είμαστε, είμαι μάλλον ε, υπεύθυνη της χώρας μου στον ΩΣΑ για την αντιμετώπιση της ε, μεταναστευτικής πολιτικής στη Βιέννη. Όλα αυτά, όλες αυτές οι θέσεις μου έδωσαν την δυνατότητα να συνεργαστώ με τους συναδέλφους από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλους εταίρους όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων είχα μία καλή εργασιακή σχέση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και διεθνή δίκτυα. Ασχολήθηκα με το θέμα ασύλου και υποστήριξης ασύλου και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣΟ. Γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά τις εργασίες, την εργασία όλων των επιμέρους, εργασίες όλων των επιμέρων ζητημάτων της ΕΑΣΟ και γνωρίζω ποιες είναι οι προκλήσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πεπισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μία στεναρή υπηρεσία ασύλου για να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις και να φτάσει σε μία ενδυναμωμένη συνεργασία στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Και εδώ θα εστιάσω την προσοχή μου αν είμαι πραγματικά, γίνω πραγματικά η εκτελεστική διευθύντρια της ΕΑΣΟ. Χρειάζεται ένα κοινό σύστημα ασύλου και γι' αυτό ε, είναι ζωτική σημασία αυτό το κοινό πλαίσιο συνεργασία. αν θέλουμε να προωθήσουμε την αλληλεγγύη, την αμοιβαία συνεργασία και την κατανόηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα κατάρτισης, δεξιότητες και σύγκληση στις διαδικασίες ε, χορήγησης ασύλου. Αυτό θα είναι και το ζωτικό έργο του οργανισμού το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου δεν καθίσταται δυνατό χωρίς να υπάρχει μία αυτόνομη ε, ροή πληροφοριών σε σχέση με τις χώρες προέλευσης καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Γι' αυτό σε εκτελεστική διευθύντρια θα ε, προωθήσω τα ζητήματα ανάλυσης ε, και επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, πολλά, ε, μάλλον μερικά κράτη που αντιμετωπίζουν οξύ ζήτημα λόγω της προσέλευσης και γι' αυτό η ΕΑΣΟ θα συνεργαστεί στενά με αυτά τα κράτη και με τους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους χρήζοντες προστασία. Θα θέλαμε να έχουμε μέσα στήριξη σε hot spots, σημεία υποδοχής και για την και, για την, στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνει είτε επαναπατρισμός είτε εσωτερική μεταφορά. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της εντολής της ΕΑΣΟ. Κατά την άποψή μου, η νέα ανασυγκρότηση της ΕΑΣΟ ήταν θετική από πολλές πλευρές. Θεωρώ ότι η διάρθρωση της οργάνωσης θα αντικατοπτρίσει τα νέα ζήτηματα και προκλήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε νέες ευθύνες μέσα στα πλαίσια της πλήρους λειτουργίας του οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατάφερε να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του για την επόμενη περίοδο, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να συνεργαστούμε και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχτεί την απαλλαγή για την ΕΑΣΟ για το 2017. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο θα πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό την επιμελητιακή βοήθεια και τους ανθρώπινους πόρους για να συμβαδίσει με τη νέα ατζέντα για την μετανάστευση με φάση τα συμπεράσματα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό μπορεί να γίνει αν συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, ο εκτελεστικός διευθύντης μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει μια ε, στρατηγική θεώρηση της ΕΑΣΟ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε μέσα και για την ΕΑΣΟ. Γι' αυτό ο εκτελεστικός ε, διευθυντής θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους υπαλλήλους, τους ανώτερους υπαλλήλους, μέσα στα πλαίσια ενός πολύ καλού εργασιακού πλαισίου. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ε, ε, ΛΥΜΠΕ, ο εκτελεστικός διευθυντής ε, της ΕΑΣΟ, είναι μια νέα πρόκληση και αυτό θα αφορά και τη δική μου σταδιοδρομία γιατί ασχολήθηκα με τη μετανάστευση και το άσυλο σε όλη την επαγγελματική μου πορεία. Υπάρχουν πολύ σοβαρές προκλήσεις ενώπιόν μας, αλλά είμαι πεπισμένη ότι από κοινού και με κοινή συνεργασία θα τα καταφέρουμε. Αυτό αφορά και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα υπάρχει κοινή θεώρηση και αμοιβαία κατανόηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you. You αυτό είναι σπάνιο, λέει ο Πρόεδρος. Στο Στρασβούργο Δευτέρα βράδυ χειροκρότημα είναι σπάνιο. Πολύ καλή αρχή. Ευχαριστούμε κυρία Γκριγκόρη. Ας ακούσουμε τώρα τα μέλη. Ξεκινώντας από τον κύριο Νίντα Μιούλα, ο οποίος εργάστηκε στο φάκελο αυτό. Πίτερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία για την εισήγησή της, την παρουσίασή της. Νομίζω ότι μετά από κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια και μήνες η ΕΑΣΟ αναδύεται ξανά με νέα δυναμικότητα και νέες δραστηριότητες. Είναι ε, μια, ένας από τους σημαντικούς θεσμούς του κοινού συστήματος ασύλου. Δεν μιλούμε μόνο πλέον για την διαχείριση και άμυνα των συνόρων που είναι σημαντικά, αλλά και για το πολύ σημαντικό πρόβλημα του πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ε, το προσφυγικό ε, θέμα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Λυπούμε ιδιαίτερα που το Συμβούλιο δεν κατάφερε να βρει μια λέση. Θα θυμάστε ίσως ότι είχαμε μια μεταβατική προσωρινή συμφωνία του Ιούλιο του 2017 με την ε, Μαλτέζικη Προεδρία και δύο χρόνια σχεδόν αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ντροπή που το Συμβούλιο δεν έκανε τίποτα. Και έχω κουραστεί να ακούω τη μία μετά την άλλη από τις Προεδρίες να λένε ότι δεν, δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα, είναι καθήκον του Συμβουλίου ώστε να γίνει ο θεσμός αυτός ενεργό κομμάτι του κοινού συστήματος ασύλου. Στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια η Άσο είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρει να εκτελέσει τα καθήκοντά της, αλλά θα πρέπει να γίνει ακριβώς οργανικά μέλος του Ευρωπαϊκού Αυτού Κοινού συστήματο Ασύλου. Εγώ σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Οι συντονιστέ, η κυρία Μέτσολα, Σίπολα, η κυρία Μέτσολα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Γκρεγόρη. Ε, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον ε, μεταβατικό αναπληρωτή κύριο Αντού που βρίσκεται εδώ σήμερα, που ηγείται του οργανισμού σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή που δυστυχώς η προσοχή επί του οργανισμού δεν ήταν θετική ή κολακευτική. Εμείς πάντοτε προσπαθούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο οργανισμός αυτός να ε, λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συμφωνώ με τον κύριο Νίτα Μίλα ε, στην απογοήτευση που εκφράζουμε σχετικά με την έλλειψη ανάληψης δράσης ή πρωτοβουλίας από το Συμβούλιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουν όλοι οι φορείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εννοεί αυτά που λέει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Χρειάζεται να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Εγώ σας εύχομαι πολύ και καλή επιτυχία στο νέο ρόλο σας, στα νέα σας καθήκοντα κυρία Γκριγόρη, για την πρόσφατη υποστήριξη που έχει δοθεί σε κάποιες ε, δράσεις, δραστηριότητες ε, εκφορτώσεων σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ο οργανισμός τι θα είχε να πει για τέτοιο είδους ad hoc υποστήριξη και πώς στο μέλλον μπορούμε να υποστηρίξουμε έναν βιώσιμο για να μην πω μόνιμο μηχανισμό στήριξης. Ευχαριστούμε Ρομπέρτα. Μπίργκετ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με ένα σύντομο σχόλιο. Ο κύριος Νίντα μου είπε ότι ήδη το 17 είχαμε μια μεταβατική συμφωνία, όμως ούτε τότε δεν είχε καταφέρει το Συμβούλιο να τοποθετηθεί με σαφήνεια επί του συστήματος ασύλου. Και θυμάμαι τότε ότι μετά την απόφαση αυτή, τη συμφωνία αυτή, το Σαββατοκύριακο, είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα ενός πολιτικού ηγέτη που έλεγε ότι θα πρέπει οι ηγέτες των εθνικών κυβερνήσεων έχουν περισσότερη, περισσότερες αρμοδιότητες γιατί μόνο αυτοί μπορούν να λάβουν ταχύες αποφάσεις. Το οποίο μου θυμίζει το θέμα των ημερών που είναι το καρναβάλι. Το κοινοβούλιο από ό,τι φαίνεται λαμβάνει ταχύτερα αποφάσεις παρά τις πολυάριθμες πολιτικές μας ομάδες. Μάλλον αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Ρωϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι η γενικού σχολείου Ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς το ρόλο σας, καθότι ακόμα περιμένουμε μια κοινή θέση, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Αυτό πώς θα επηρεάσει τη δουλειά σας. Πώς εσείς μπορείτε να προετοιμαστείτε για τη στιγμή κατά την οποία θα έχουμε επιτέλους το κοινό σύστημα. Πώς βλέπετε εσείς τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσετε, καθότι η κατάσταση στη μετανάστευση και στο άσυλο αλλάζει διαρκώς. Και στο παρελθόν συνέβαινε αυτό και ακόμα αλλάζει. Έχουμε νέα γεγονότα, νέες προκλήσεις, ιδιαίτερη, ιδιαίτερα πολιτικοποιημένες, πολιτικά ευαίσθητες συζητήσεις και ανταλλαγές. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η Άσο να είναι αποτελεσματική. Ακόμα και χωρίς μια σαφή τοποθέτηση και απόφαση Συμβουλίου. Ευχαριστούμε την Μπίργκη την Ναταλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εξ ονόμαστε της και της ε, Σεσίλια Βίξτοχον που δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε, που είναι ειδική εξημών για τα θέματα αυτά. Σας ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία και για τα νέα σας αυτά καθήκοντα πρόκειται να αναλάβετε που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους πολίτες, όχι ο ίδιος ο οργανισμός, αλλά όπως καταλαβαίνετε το όλο φαινόμενο, το όλο πρόβλημα. Απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία. Και συνεχίζοντας σχόλια των συναδέλφων που μίλησαν προηγουμένως ε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευση, την έντονη απογοήτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνοντας την απόλυτη αδράνεια του Συμβουλίου απέναντι στο φάκελο αυτό. Ανεξαρτήτως πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο βλέπετε ότι έχουμε επιτύχει μια συνένεση για την κατάσταση αυτή την οποία, η οποία είναι πραγματικά θλιβερή. θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου αντίθετα για την ε, άφηξή σας που ίσως να γυρνάει μια νέα σελίδα για τον οργανισμό μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Αυτό θα είναι πολύ καλό. Η ερώτηση μου λοιπόν ίσως είναι λιγότερο γενική, το πήρα αντίστροφα, ε, σχετικά με τις τελευταίες εκθέσεις για τα hot spot αντιλαμβάνεται κανείς ότι η υποδοχή των ανθρώπων αυτών την χάνει πολύ καλύτερη σε διαχείριση ότι η καταπολέμηση των ανθρεμπόρων έχει επιτέλους μπει στο θεματολόγιο των θεσμών, αλλά ότι έχουμε πολύ σοβαρές παραβιάσεις, κρούσματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κέντρα αυτά που τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. με εμπορίο ανθρώπων, με καταναγκαστική δουλειά και πολλά άλλα. Ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω αυτή την πτυχή. Εσείς έχετε φανταστεί, έχετε κάποιον, κάποια κατεύθυνση για το πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την κατέστηση αυτή και πώς θα επίσης θα μπορέσετε να διευκολύνεται την ταυτοποίηση ευάλωτων ανθρώπων και εδώ μιλώντας ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των παιδιών, των ανηλίκων που βρίσκονται μεταξύ των μεταναστών και των προσφύγων. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ Helga Stevens λέει ο πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κυρία Γκρεγόρη για την εισαγωγή της και θα ήθελα να, της, ε, να την ρωτήσω ποια, είναι η πρόθεσή της ε, σχετικά με την, ιδιαίτερα με την πολιτική για το προσωπικό. Δηλαδή πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση σε σχέση με αυτά που γινόντουσαν μέχρι εδώ. Ε, είστε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία μου, αλλά είστε και υποψήφια για, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Πώς θα αποφύγετε μια δυνητική σύγκρουση συμφερόντων. Είστε μέλος του Οικειητικού Συμβουλίου. Για τους υποψηφίους διευθυντές θα μπορούσατε να έχετε τοποθετηθεί. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο ακόμα στοιχείο. Κύριε Άινστ, σας ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρουσίασή σας και γνωρίζουμε όλοι πως η ΕΑΣΟ, πώς να το πω, έχει αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες, ακόμα περισσότερες από αυτές που είχε. Και παρατηρούμε επίσης πως στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και αλλού υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στα σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ακούμε ξανά και ξανά πως είναι μεγάλο πρόβλημα, πως πρέπει να κάνουμε κάτι, όμως θα ήθελα από εσά να μου πείτε τι συμβαίνει με το δικαίωμα διεθνούς προστασίας και ποιο ρόλο θα παίξει ε, στο έργο σας ε, ως εκτελεστική διευθύντρια της ΕΑΣΟ στο μέλλον. Με λίγα λόγια, πώς θα συνεισφέρετε έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δικαίωμα προστασίας ε, των προσφύγων και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Η Άσου λοιπόν έχει σημαντικό ρόλο εδώ. Επίσης, μου προκάλεσαν έκπληξη, αν όχι με σόκαραν αυτές οι δηλώσεις που διάβασα για τα κέντρα ελέγχου, τα ελεγχόμενα κέντρα, τα control centers. Κατά τη δική σας γνώμη, ποιο ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η ΕΑΣΟ ε, σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε απελάσεις, επιστροφές και πόσο μεγάλο μερίδιο του όγκου της δουλειά σας ε, θα καταλάβει αυτό το σκέλος. Σας ευχαριστώ. Okay, just... Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα δώσουμε και στην κυρία Γκρεγόρη 10 λεπτά χρόνο για να καταφέρει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Νομίζω πως είναι δίκαιο. Ο κύριος Τερικάμπρας έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Γκρεγόρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και που απαντήσατε εκ των προτέρων στις ερωτήσεις μας. Έχω τις εξής ερωτήσεις. Η πρώτη συνδέεται και με την ε, τελευταία ερώτηση της κυρίας Έρνστ. Εάν διοριστείτε, ναι, εκτελεστική διευθύντρια της ΕΑΣΟ, πώς θα διασφαλίσετε ότι η ΕΑΣΟ δεν θα υπερβαίνει των αρμοδιοτήτων της και του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άσυλο. Επίσης, αναφερθήκατε στα ελεγχόμενα κέντρα και πλατφόρμες διάδοση. Όμως, το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν περιλαμβάνει τέτοιες έννοιες. Πώς λοιπόν θα διασφαλίσετε ότι το έργο της ΕΑΣΟ θα είναι εντός των αρμοδιοτήτων της και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου. Έπειτα, δεύτερη ερώτηση. Με το ρόλο σας ως νέα διευθύντρια, πώς θα φροντίσετε να εξασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της ΕΑΣΟ. Και τρίτη ερώτηση. Η κοινωνία των πολιτών, με τις ε, διάφορες οργανώσεις. Πώς θα συμμετάσχει, αν θα συμμετάσχει και στην, ε, στον έλεγχο και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων της ΕΑΣΟ. Και πώς μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία με το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τερικάμπρας. Η Μάιτε, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Αυτό που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πρώτα απ' όλα να βοηθήσετε, να ενισχύσετε την αξιοπιστία του οργανισμού που σε διάφορα επίπεδα δεν έχει τη φήμη ότι είναι πολύ αποτελεσματικός λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω διαφόρων αιτιών. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία από διάφορες συναντήσεις και με διάφορους φορείς και στο πεδίο και επομένω είμαι σίγουροι ότι θα γνωρίζετε όλες τις υπηρεσίες, τα γραφεία της ΕΑΣΟ εκεί όπου επιχειρεί. Και ίσως αυτή η μεταφορά γραφείων, για, για παράδειγμα στο κέντρο της Μόρια, από την οποία επέστρεψα προχθές, στην ουσία μιλούμε για ένα άθλιο μπούνκερ. Ε, και φαντάζομαι ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα όταν αναφέρεστε σε, σε προβλήματα είναι πού βρίσκονται αυτοί οι χώροι. Πώς μπορεί να συνεργαστεί κανείς με τα γραφεία αυτά, με τις υπηρεσίες αυτές. Για τα μαύρα αυτά σημεία και πρέπει να σας πω ότι η Μόρια είναι πραγματικά δηλαδή απαράδεκτη. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και με την έλευση Αφγανών στα ελληνικά νησιά για παράδειγμα. Πώς θεωρείτε όταν δεν μπορούν να επιστραφούν στο Αφγανιστάν Πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση που δεν θα επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων αυτών, ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα, για παράδειγμα. Τα παιδιά, τους ανελίκους, τους απάτριδες που ε, έρχονται στη ζωή σε διάφορα σημεία όλης αυτής της περιπέτειας, της πορείας των ανθρώπων αυτών. Επομένως θέλω να πω ότι τα προβλήματα πεδίου και όχι υψηλού επίπεδου είναι τα πιο σημαντικά. Η έλλειψη του προσωπικού. Πραγματικά ε, πρέπει να μας το εξηγήσετε, να μας το περιγράψετε γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε τον οργανισμό. Ευχαριστώ. Νομίζω πω αυτή ήταν πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ήθελα και εγώ να την ε, κάνω. Αυτό το παράδειγμα που μας έδωσε η Μάιτε για τη Δυτική Μεσόγειο είναι πάρα πολύ ενδεικτικό νομίζω. Πώς ε, μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις προσδοκίες των πολιτών και ε, να τους ενημερώσετε για το τι ακριβώς κάνει η ΆΣΟ, ποιες αρμοδιότητες έχει. Παρατηρώ πως υπάρχει μία ένα πρόβλημα στο, στην κατανόηση των πολιτών σχετικά με το τι κάνει η υπηρεσία σας. Και νομίζω πως ε, αυτή θα είναι μία από τις ε, πρώτες ε, μεθοδευτές σας. Η Άννα έχει τώρα το λόγο. Κυρία Γκρεγόρη, και εγώ όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη στο έργο σας, διότι είναι πολύ δύσκολο σίγουρα. Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω έχει ήδη γίνει από τους συναδέλφους. Δηλαδή, πώς ε, βλέπετε το ρόλο της ΕΑΣΟ στις ε, διάφορες ε, διαδικασίες απέλασης και επιστροφής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι που επιστρέφονται δεν προέρχονται από ασφαλείς χώρες, όπως το Αφγανιστάν, για παράδειγμα. Ε, βέβαια, η ΕΑΣΟ θα είχε διαφορετικό ρόλο σε όλα αυτά, εάν υπήρχαν νόμες μεταναστευτικές οδοί και δεν επιτρέπαμε στους διακινητές και στους ε, ελευθερούς να ε, διαχειρίζονται την ε, μετανάστευση. Έχετε πίγνωση της πραγματικότητας ή όχι. Επίσης, η υπηρεσία σας έχει έδρα τη Μάλτα. Η Μάλτα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Πρόκειται για ένα κράτος μέλος το του οποίου η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα παράνομης έκδοσης θεωρήσεων σε παράτυπους μετανάστες από την Αλγερία, από τη Βόρεια Αφρική κτλ. Τα διαβάζουμε αυτά στα μέσα ενημέρωσης. Και ορισμένοι από εμάς μάλιστα έχουν υποβάλει και ε, γραπτές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγνοούμαστε όμως. Μας αγνοεί μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς ε, τι πρόθεση έχετε, να συνεχίσετε να αγνοείτε όλα αυτά, να στουρθοκαμιλίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος? Αυτές ήταν οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Σίγουρα ο ρόλος σας έχει πάρα πολλές προκλήσεις και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο και το χρόνο να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων όσο το δυνατόν ε, πιο Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μπω στην ουσία για να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί πρόκειται για ζητήματα τα οποία, πώς να το πω, είναι προβληματικά, είναι νευραλγικά σημεία και όχι μόνο για την άσο. Αυτό αυτό το πάγωμα του σχεδίου κανονισμού για την ΕΑΣΟ σίγουρα δεν μας διευκολύνει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω στις ερωτήσεις σας με τη σειρά που εκείνες ετέθησαν και ελπίζω να καταφέρω να τις ομαδοποιήσω κάπως. Όμως, να ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Νίτερ του εισηγητή για την ΕΑΣΟ. Καταρχάς να πω πως είναι πολύ σημαντική η θέση σας ως ε, εισηγητή ε, γιατί γνωρίζετε καλύτερα το θέμα βέβαια. Σίγουρα, αν δούμε όλο το θέμα σφαιρικά ως ε, ένα σύνολο, θα ήταν καλύτερα. Όμως, έτσι όπως περιγράφεται την κατάσταση, με το αδιέξοδο μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου πραγματικά είναι κρίμα να μην ε, έχει σημειωθεί καμία πρόοδος ε, για την ΕΑΣΟ, διότι αυτό θα μας έδινε πρόσθετες δυνατότητες. Θα είχαμε ε, επιπλέον στήριξη και θα μπορούσε με την στήριξη αυτή η ΕΑΣΟ να βοηθήσει εκείνους που χρειάζονται προστασία. Η υπηρεσία μας αυτή τη στιγμή έχει την εντολή να στηρίζει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαδικασία ασύλου. Άρα λοιπόν πρώτα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, εφαρμογή του ε, κοινού συστήματος ασύλου και γι' αυτό πρέπει να δούμε πως ε, χρειάζεται δημιουργία εργαλείων για το, την εκείνη νομοθεσία περί ασύλου, υποδομών, κατάρτιση προσωπικού και αυτό φυσικά δεν γίνεται χωρίς μια πληρέστερη εντολή της ε, ΕΑΣΟ, η οποία φυσικά θα βοηθούσε έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε ακόμα καλύτερα τα κράτη-μέλη και να αποφύγουμε ε, τις ε, καθυστερήσεις, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στην αντιμετώπιση κρίσεων. Δυστυχώς και εμείς στην ΕΑΣΟ το θεωρούμε λυπηρό. Ελπίζουμε όμως μια διευρυμένη εντολή να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον για να μας βοηθήσει. Μετά, η κυρία Μετσόλα αναφέρθηκε στα προσωρινά μέτρα και στις ε, ad hoc επιχειρήσεις αποβίβασης ε, ανθρώπων. Η Άσο πράγματι πρόσφερε τη στήριξή της στα κρατημέλη που την χρειάζονταν, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Μάλτα. Όμως, εμείς εξαρτώμαστε από την ε, συγκατάθεση των ε, κρατών μελών. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν συμφωνήσουν. Είχαμε λοιπόν ε, την περίπτωση της Μεσίνας στην Ιταλία, όπου η ΕΑΣΟ είχε στείλει εμπειρογνώμονες, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, βοήθησε στην ε, μεταφορά της πληροφορίας, στην καταγραφή, τη συνεντεύξεις ε, των ε, μεταναστών εκ μέρους του κράτους μέλους. Και φυσικά εδώ είδαμε πόσο σημαντικό ήταν να υπάρχει συντονισμός επιτόπου. Διότι με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποκομίσουν μία ρεαλιστική εικόνα του τι συμβαίνει. Και αυτό βοηθά και για το μέλλον. Φυσικά τα προσωρινά μέτρα δεν μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν ένα βιώσιμο σύστημα για το μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε βάση στο ε, κράτος μέλος άφηξης. Και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς αυτά τα προσωρινά μέτρα μπορούν να μετατραπούν σε ένα βιώσιμο σύστημα και για μετεγκατάσταση. Ελπίζω να αποτελέσουμε το καλό παράδειγμα και να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτά τα προσωρινά μέτρα να γίνουν ένα πλήρες σύστημα στήριξης. Έπειτα. Η κυρία Ζίπελ έκανε μια ερώτηση σχετικά με την διευρυμένη εντολή για την ΕΑΣΟ. Και πώς μπορεί η ΕΑΣΟ να συνεχίσει χωρίς αυτήν. Να πω καταρχάς ότι... Καταρχάς, εάν η ΕΑΣΟ λάβει επιπλέον χρηματοδότηση, θα έχει και περισσότερες δυνατότητες να απασχολήσει μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, για παράδειγμα. Στο πούμε ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 212 υπαλλήλου στη Μάλτα και 170 στην Ελλάδα, σε διάφορες επιχειρήσεις. Και στην Ιταλία έχουμε άλλους 170, 40 ε, επίσης στην Κύπρο, με μια διευρυμένη εντολή θα υπήρχε μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά του ανθρώπινου πόρου. Η Κομισιόν βέβαια πρότεινε να αυξηθεί ο αριθμό του προσωπικού στη Μάλτα στου 500 και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός από τα 69 εκατομμύρια τώρα στα 300 εκατομμύρια και αργότερα σε βάθος χρόνου με περισσότερη χρηματοδότηση μπορούμε φυσικά να κάνουμε και περισσότερα. Βέβαια, μέχρι τη στιγμή εκείνη η Άσο θα προσπαθήσει να προσλάβει όσο το δυνατόν ε, περισσότερο καλά καταρτισμένο προσωπικό. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τον υποστηρικτικό μας ρόλο στα κράτη-μέλη. Μετά, η κυρία Γκρίσπεκ ε, έκανα μια ερώτηση για την έκθεση σχετικά με τα hot spots. Και σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις εκεί. Σίγουρα είναι μέρος της, ε, των ομορδιοτήτων της ΕΑΣΟ, είναι μέρο μέρος του συστήματος ε, ασύλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η ΕΑΣΟ θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις ε, κυριότερες προκλήσεις που ήδη αναφέρεται. Πρέπει καταρχάς ε, να αποτελεί κύριο μέλημά μας το... τα παιδιά, η καταπολέμηση της ε, έμφυλης Χρειαζόμαστε λοιπόν την κατάλληλη κατάρτιση, υποστηρικτικά εργαλεία, ενημέρωση και να παρέχουμε βοήθεια στα κράτη-μέλη στους τομείς αυτούς. Αυτή όμως είναι μια προσπάθεια που γίνεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και φυσικά η συνεργασία μας με την υπηρεσία αυτή όλο ένα και βελτιώνεται. Και πρέπει να πω εδώ ότι η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια είναι πάρα πολύ καλή και υπάρχουν ορισμένοι τομείς ε, στους οποίους αριστεύουμε. Το 2018 η ΆΣΟ μαζί με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ανέπτυξε νέα εργαλεία καθοδήγησης για τις συνθήκες υποδοχής ασυνόδευτων παιδιών. Εξέδωσε και έναν οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση των ε, μέρους περιπτώσεων και νομίζω πως ε, αυτό δείχνει και την καλή συνεργασία που έχουμε με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και το 2019 εξέδωσε έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών για ε, το, τους ασυνόδευτους ανήλικους. Επίσης, η ΆΣΟ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο για την προστασία των ευάλωτων προσώπων στην διαδικασία χορήγησης ασύλου και νομίζω πως αυτό είναι ένα πολύ θετικό ε, στοιχείο, το οποίο φυσικά και θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Τώρα σε ό,τι την κοινωνία των πολιτών και το ρόλο της. Πράγματι, ισχύει αυτό που είπατε. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο κανονισμό, η ΕΑΣΟ προσπαθεί να προσελκύσει την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα ασύλου. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της ε, πολιτικής νομοθεσίας, της υλοποίηση ε, σχετικών μέτρων και όπως είπατε και εσείς, το Συμβουλευτικό Φόρουμ ε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός με πάνω από 150 μέλη. Και εκεί γίνεται πολύ σημαντική δουλειά χωρίζεται σε τρεις τομείς δραστηριοτήτων. Πρώτον υπάρχει η ετήσια ολομέλεια και οι τακτικές συνεδριάσεις του φόρουμ. Ε, υπάρχει η ηλεκτρονική διαδικασία διαβούλευσης για τα κυριότερα έγγραφα με τα οποία ασχολείται η ΕΑΣΟ και ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΕΑΣΟ, όπως για παράδειγμα ε, το δίκτυο εμπειρογνωμόνων. Όπως σας είπα, είναι ενεξελίξει το όλο πρόγραμμα και προσπαθούμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας με την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει το Συμβουλευτικό Φόρουμ και ελπίζουμε ε, με τη διευρυμένη εντολή της νέας υπηρεσίας να ε, ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Τώρα, τι γίνεται επιτόπου, τι γίνεται με τις ε, συνθήκες στα hot spot και τα κέντρα υποδοχής. Νομίζω πως ε, όλοι γνωρίζουμε τις ε, δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα αυτά, οι οποίες σίγουρα αποτελούν μεγάλη πρόκληση και για εμάς Υπάρχουν πολλοί εμπειρογνώμονε από κράτη-μέλη που εργάζονται σε αυτά τα κέντρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασφαλίζονται οι κατάλληλε ε, συνθήκε στα κέντρα αυτά. Η ΆΣΟ αυτή τη στιγμή έχει υποστηρικτικό ρόλο όπου μπορεί, πάντα σύμφωνα με την εντολή της. Διότι τα κέντρα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και ο ρόλος μας είναι να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες και τα παιδιά, ε, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τις αρχές, έτσι ώστε η διαδικασία ασύλου να είναι σύντομη και ασφαλής, για να μην μένει ο κόσμος πολύ σε αυτά τα μέρη. Όμως ε, θεωρώ πως σίγουρα υπάρχει πολύ καλός ε, συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων και ο ρόλος της ΕΑΣΟ εδώ είναι να βοηθάσω το δυνατόν ε, περισσότερο και καλύτερα τις ε, αρχές ε, για την βελτίωση των συνθήκων στα κέντρα αυτά. Και φτάνουμε στην ερώτηση του κυρίου Μωράης. Ποιε είναι οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΟ. Νομίζω πως είναι σαφές ε, πως οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΟ είναι αρκετά περιορισμένες εδώ. Εδώ πρακτικά η ΆΣΟ μπορεί να ενισχύσει και να βελτιώσει τις, ε, τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ε, στην ε, παρακολούθηση και τον έλεγχο του, της διαδικασίας χορήγησης ασύλου η ΆΣΟ παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και αναπτύσσει νέες προσεγγίσεις μαζί με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Όλα αυτά μπορούν φυσικά να βοηθήσουν, όμως είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει. Συγγνώμη που σας διακόπτω, ε, διακόπτω λέει ο πρόεδρο, ε, δεν έχει να κάνει με προσδοκίες. Ε, είναι... Έχει να κάνει με το τι περιμένουμε από εσά. Όμω, επειδή τελειώνει ο χρόνος, και να σας ζητήσω ξανά συγγνώμη που σας διέκοψα, υπάρχουν ερωτήσεις που έχουν μείνει αναπάντητες σχετικά με την επιστροφή και τον επαναπατρισμό μεταναστών. Η Άννα Γκόμες νομίζω την ε, έκανε, οπότε θα ήθελα να απαντήσετε αν μπορείτε. international protection. Και θέματα διεθνούς ε, προστασίας, ναι, σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο. Ναι, επαναπατρισμός ε, και επιστροφές δύναμη του κοινοτικού δικαίου και του ε, δικαίου περί διεθνούς προστασίας η ΆΣΟ δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιστροφών. ως προς τη λήξη της διαδικασίας ασύλου και επαναπατρισμού. Αυτό είναι θέμα ECBG ή Frontex. Η ΆΣΟ δεν έχει εντολή για τους επαναπατρισμούς. Η ΆΣΟ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στη διαδικασία χορήγησης ασύλου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τα κράτη-μέλη έχουν το σωστό, τη σωστή πλαισίωση για τον επαναπατρισμό βεβαίως και με βάση τα δεδομένα της Frontex ως προς τον επαναπατρισμό στη χώρα προέλευσης. Αυτό θα πρέπει να το διασαφηνίσουμε γιατί ο κόσμος θα πρέπει να ε, κατανοήσει ποιο είναι και οι περιορισμοί, περιορισμοί της ΕΑΖΟ. Αυτό ήταν και ένα άλλο ερώτημα της κυρίας Κόμες. Ε, είσαστε όλοι ικανοποιημένοι. Υπάρχουν ε, επιπρόσθετες ερωτήσεις. Ξέρω ότι αυτή η διαδικασία δεν ε, ε, ολοκληρώνεται πάντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία ε, Γκρεγόρη για την παρουσία της. Ευχαριστώ και τα μέλη για τις ερωτήσεις. Και τώρα έχουμε τη σύσταση ΛΥΜΠΕ για μία γνωμοδότηση. Αυτό θα αποφασιστεί από τους συντονιστές με γραπτή διαδικασία. Εάν συμφωνείτε όλοι, ευχαριστώ την κυρία Γκρεγόρη για την παρουσίασή της και για την παρουσία σας στο Στρασβούργο τη Δευτέρα το απόγευμα. Ευχαριστώ και τις ερωτήσεις των μελών σας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και αυτό αφορά και το προσωπικό σας φυσικά. Ευχαριστούμε. So, colleagues... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε τώρα στην ε, πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Um, Ξέρω ότι είναι κουραστική διαδικασία. Δευτέρα βράδυ στο Στρασβούργο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε το θέμα της ανταλλαγής απόψεων σχέση με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Όπως ξέρετε πρόκειται για μέτρα καταπολέμησης της προπαγάνδας και άρση και απόσυρση του περιεχομένου. Ο κύριος Ντάλτον δεν είναι εδώ. Η Helga Στίβενς τον αντικαθιστά. Ωραία. Έχουμε τουλάχιστον ένα-δύο σκιώδεις. Θέλετε να μιλήσετε ως προς τις τροπολογίες. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί ο κύριος ε, Ντάλτον δεν είναι παρόν ε, σήμερα, τον αντικαθιστώ, αλλά θα σας ε, διαβάσω τις δικές του σημειώσεις. Ζητώ συγγνώμη ε, για την απουσία του. Από την τελευταία μας συζήτηση στην Επιτροπή είχαμε πάνω από 700 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Ε, είναι μεγάλη πρόκληση λοιπόν να ευρεθούν συμβιβασμοί, όμως δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επί του θέματος ε, από το Κοινοβούλιο. Ως εισηγητής θέλω να φτάσουμε στην ευρύτερη δυνατή συμφωνία πριν από την ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε μία ε, ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε την δεύτερη συνάντηση σκιωδών ε, την προηγούμενη εβδομάδα και αύριο την επόμενη. Και προβλέπονται και άλλες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα. Οι 700 τροπολογίες που υποβλήθηκαν δείχνουν απόκληση απόψεων σε ορισμένα βασικά στοιχεία της πρότασης. Άρση, θέματα άρσης και αφαίρεσης περιεχομένου, αλλά υπάρχουν και κοινά σημεία που θα αποτελέσουν βάση της συμφωνίας. Ε, όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να είναι στοχοθετημένη η πρόταση σε σχέση με τη διάδοση ε, συγκεκριμένων ε, αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου που θα πρέπει να αποσυρθούν. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνεται και με τις υπηρεσίες νέφους που δεν μπορούν να αφαιρέσουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορεί πολλές φορές να χρησιμοποιήσουν λάθος αυτά τα δεδομένα σε επίπεδο πρώτης επαφής. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που αφορά ε, εξαιρέσεις. Θεωρούμε ότι οι ΜΜΕ δεν θα πρέπει να έχουν μεγάλο φόρτο λόγω του κανονισμού, αλλά ανησυχώ όταν μιλάμε για κατόφλια τα οποία δείχνουν ε, μεγάλη νομοθετική αποτυχία κατά την απόψή μου. Θα πρέπει να είναι αναλογικός ο κανονισμός και να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους. Ως προς τον ορισμό τρομοκρατικού περιεχομένου, αυτός ο τομέας χρήζει περαιτέρω συζήτησης για να είμαστε σωστοί ε, ως προς τις διατυπώσεις μας δεν θέλουμε να κινηθούμε πέραν της οδηγίας περί αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Μία από τις βασικές μου ανησυχίες και ένα βασικό μου μέλημα που συμμερίζονται και τα μέλη είναι ότι τα θέματα περιορισμένης, περιορισμού ευθυνών ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα πρέπει να υποσκάπτονται και δεν θα πρέπει να αφήσουμε παραθυράκια σε αυτό το κανονισμό. Χρειάζονται περαιτέρω συζητήσει σε σχέση με τη διατύπωση του άρθρου 6 αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμφωνίες. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εθελούσια μέτρα θεωρώ ότι οι κινήσεις μας για τα εντάλματα απόσυρσης θα πρέπει να μας, ε, να μας απασχολήσουμε στα πλαίσια και του χρονικού αυτού προσδιορισμού. Υπάρχουν και οι επιπτώσεις της ε, ΜΜΕ. Μεγάλος φόρτος δηλαδή. Και γνωρίζω ότι δεν θα πρέπει να θα πρέπει να υπάρξει αναχέτηση του, των καταχωρήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου και γι' αυτό χρειάζονται σαφείς κανόνες πριν φτάσουμε σε ένα συμβασμό. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε ε, διασυνοριακά εντάλματα άρσης αλλά με ρήτρες διασφάλισης που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του κανονισμού. Σε σχέση με το άρθρο 5 της εκούσιες αναπομπές υπάρχουν υπάρχουν, ε, υπάρχουν ε, αποκλήσεις σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης και πληροφορίες, αν και υπάρχουν ε, επιχειρήματα σε σχέση με το κατά πόσο είναι μέσο συνεργασίες για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Βεβαίως, οι κυρώσεις είναι ένα βασικό θέμα αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση σε σχέση με ένα ευέλικτο σύστημα κυρώσεων που θα λαμβάνει υπόψη και ελαφρυντικά. Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις όταν κανείς συστηματικά δεν ανταποκρίνεται. Αυτός θα πρέπει να είναι και ένας, ε, αυτή θα πρέπει να είναι και μία διαδικασία που αφορά ε, μία ε, όχι και τόσο αμετροεπή προσέγγιση έτσι ώστε να μην αφαιρείται κάθε περιεχόμενο. Η ομάδα μου θα παρακολουθήσει την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και θα παρακολουθήσω την όλη διαδικασία αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ. Αυτή η ομάδα στην οποία αναφερθήκατε έχει και άλλα μέλη, πρώτα ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε Χέλγα Ευχαριστούμε τους ε, συναδέλφους που έμειναν, γιατί πολλοί άλλοι δεν κατάφεραν να είναι εδώ μέχρι αυτήν την ώρα. Ρομπέρτα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε που το καλύπτεις ε, το θέμα. Είναι σημαντικός ο φάκελος. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την κυρία Ντάτη πράγματι για να εξηγήσω τις προτεραιότητες της δικής μας ομάδας σε αυτό το φάκελο. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και προσπαθώντας να βρούμε συμβαστικές λύσεις σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, σημαντικές διαφορές και ας είμαστε δίκαιοι οι κοινέ γραμμές σε αυτόν εδώ το φάκελο είναι κάτι δύσκολο. Εδώ μιλούμε για έναν κανονισμό για την ενίσχυση της ε, καταπολέμησης της online παρουσίας τρομοκρατικών οργανώσεων. Για όσους δεν πιστεύουν στην αξία της πρότασης αυτής, πρέπει να θυμόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι μία από τις βασικότερες οδούς ριζοσπαστικοποίησης. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποστείλουμε κάποιο μήνυμα αδυναμίας στις διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και τους προπαγανδιστές τους. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες και να εργαστούμε από κοινού για έναν πιο ισχυρό κανονισμό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το τρομοκρατικό περιεχόμενο του διαδικτύου. Η κυρία Ντάτη δεν μπορεί να δεχθεί λοιπόν διάφορες μερικές μάλλον από τις τροπολογίες οι οποίες αποδυναμώνουν τις διατάξεις του κανονισμού. Χρειαζόμαστε προδραστικά μέτρα δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή είναι η γραμμή που είχε εξάλλου υιοθετήσει και το Συμβουλίο και η Επιτροπή. Δεν πρέπει λοιπόν να αποδυναμωθεί ο κανονισμό αυτό και ελπίζουμε ότι η συζήτηση που θα έχουμε τι επόμενε μέρε θα είναι επικοδομητική προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μα να ψηφίσουμε το τέλος της, στο τέλο τη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε, Ρομπέρτα και η Μπίργκετ αντικαθιστά τον Τζο Βάιντεν Χόλσερ. Οπότε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρωτού πάω στις λεπτομέρειες τροπολογιών να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Τίνουμε να θεωρούμε ότι κάθε φορά που θα βρούμε μια απόφαση επί φακέλου θα επιλύσουμε την όλη κατάσταση. Αυτό δεν είναι αληθές. Μιλώντας για το διαδίκτυο και την ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο ισχυρές προσπάθειες προκειμένου να αντισταθμίσουμε τα τρομοκρατικά μηνύματα στο διαδίκτυο. Απλώς η διαγραφή κάποιων από αυτά δεν θα βοηθήσει, φοβούμε. Και νομίζω ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια σε αυτά τα εξισορροπητικά αν θέλετε μηνύματα. Θα συνεχίσω στα γερμανικά καθότι έχω τις σημειώσεις μπροστά μου στα γερμανικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς σχετικά με το ποιος είναι ο στόχος αυτής της ε, πρότασης. Η πρόταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ο στόχος πρέπει να είναι η απομάκρυνση παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου. Και επίσης ε, θα πρέπει καταρχάς να διευκρινίσουμε τι συνιστά παράνομο περιεχόμενο. Χρειάζεται λοιπόν ένα σαφής ε, ορισμός του παράνομου περιεχομένου έτσι ώστε να αποφευθούν παρανοήσεις ε, και παρεξηγήσεις που θα οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα το, τη διαγραφή παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου, είναι επίσης σαφές ότι όταν χαρακτηρίζεται ένα τέτοιο περιεχόμενο ως ε, ακατάλληλο, ως παράνομο, θα πρέπει αυτόματα να διαγράφεται. Οι αρμόδιες αρχές, εάν δεν αξιολογούν ένα, ε, κάτι, ε, κάποιο περιεχόμενο ως παράνομο, τότε θα πρέπει να μεταδίδεται η απόφαση αυτή ε, στην ε, υπηρεσία που το φιλοξενεί διαδικτυακά, έτσι ώστε να προχωρήσει και εκείνη στη δική, στη της αξιολόγηση και όχι να ε, παρεμβαίνουν οι αστυνομικές αρχές. Ο πάροχος λοιπόν υπηρεσιών θα πρέπει να έχει λόγο στο περιεχόμενο, στη διαγραφή του ή όχι. Μετά. Δεν θεωρούμε πως η νομική βάση είναι η κατάλληλη και μάλιστα το θεωρούμε κάπως περίεργο, διότι η νομική βάση για τον κανονισμό αυτό ε, κινείται στο πλαίσιο της ε, ενιαίας αγοράς και θεωρούμε λοιπόν λάθος να χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό. Όμως, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει τον, ε, την νομική βάση για την ε, νέα αγορά και την χρησιμοποιεί ως βάση για την επεξεργασία ε, του κανονισμού για το παράνομο ή το για τρομοκρατία περιεχόμενο, τότε αναρωτιέμαι γιατί δεν έλαβε υπόψη την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι η στην οδηγία αυτή αναφέρεται ότι οι πλατφόρμες φιλοξενής, οι δηλαδή υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να ε, θεωρούνται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που φιλοξενούν και βέβαια ε, σίγουρα βρισκόμαστε προ ευρωεκλογών δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το επόμενο κοινοβούλιο να μην έρθει στην άσχημη θέση να αποφασίσει για το αν θα πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο δικαστήριο. Γεγονό είναι ότι το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο δεν ανήκει στο διαδίκτυο, πρέπει να απομακρύνεται. Γι' αυτό όμω θα χρειαστεί και η ύπαρξη τη κατάλληλη νομική βάση, την οποία πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων αποφασίσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η σκιώδη των ε, Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και την Επιτροπή για την πρόταση. Θεωρούμε ότι ο εισηγητής έχει κατέβαλε σημαντική προσπάθεια σε κάποια από τα ζητήματα ιδιαίτερα στην προσπάθεια της αντιμετώπισης ε, των μηνυμάτων στο διαδίκτυο ε, ιδιαίτερα αυτών που απευθύνονται στο σύνολο του κοινού και γίνεται μια παραπομπή στην οδηγία. Τα άρθρα 5 και 7 της οδηγίας ε, ενέχουν διατάξεις ε, που θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν να ε, παράσχουν ένα πλαίσιο για την προσπάθεια αυτή. Και αυτό προκειμένου να αποφύγουμε επικαλύψεις, καθυστερήσεις και να είναι η προσπάθειά μας πιο αποτελεσματική όπως επιθυμούμε. Ωστόσο υπάρχουν σοβαρά πολιτικά προβλήματα και θα έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να τα επιλύσουμε. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε διότι η πρόταση ε, συμπεριλαμβάνει στοιχεία που δεν έχει επαρκή, που δεν έχουν ε, ε, επαρκή ασφάλεια δικαίου και ιδιαίτερα το πλαίσιο των κυρώσεων. Ε, υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Εγώ σκιώδης θα επιχειρήσω να παρουσιάσω αυτά ε, που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα ώστε να εξευρεθεί η συνένεση. Όταν μιλούμε για προδραστικά μέτρα για παράδειγμα, έτσι όπως ετέθη το θέμα, δεν θα έχουμε επαρκή χρόνο να έχει ασφάλεια δικαίου η πρόταση αυτή, το τμήμα αυτό της πρότασης. Θα μπορούσαν όμως αυτά τα μέτρα να είναι εθελοντικά, θα μπορούσαμε να πάμε σε μια φάση πιλωτικών δραστηριοτήτων, ώστε να επανέλθουμε με πολύ πληρέστερη ασφάλεια δικαίου και κάποια εμπειρική ε, ε, ε, κάποια στοιχεία που θα έχουμε συλλέξει σχετικά με το πώς θα λειτουργούν αυτές οι δράσεις στην πράξη, που δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσουμε λοιπόν να επεξεργαστούμε καλύτερα την πρόταση αυτή, η εθελοντικότητα και μια πιλωτική φάση σχεδίων θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Τώρα, σχετικά με την απόσυρση σε μία ώρα παράνομου περιεχομένου, καθότι μιλούμε για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας με με τους αλγορίθμους που έχουμε σήμερα, όλα αυτά είναι απολύτως αδυνατά. Και το τρίτο στοιχείο που είναι θεμελιώδες και επί του οποίου θα μπορούσαμε να στηριχτούμε περισσότερο στην πρόταση θεωρούμε είναι η δικαστική αρμοδιότητα. Η αρμόδια αρχή θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο στην χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Ο δικαστικός έλεγχος είναι μόνο αυτός ο οποίος θα ελέγχει σχετικά με οποιαδήποτε παρατυπία ή απόκληση από τους στόχους της πρότασης που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν σημειωθεί κάποιες ε, πρόοδοι από πλευράς του εισηγητή του κ. Ντάλτον, αλλά η ασφάλεια δικαίου σε ένα θέμα τόσο λεπτό, τόσο τεχνολογικά απαιτητικό, είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Επομένως, επαναλαμβάνω, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα θελαντικό μέσο που να είναι μετρήσιμο και να μπορέσουμε να υπολογίζουμε κατά πόσον έχουμε ήδη τα στοιχεία ώστε να μπούμε σε μια εφαρμοστική φάση στην, στην ερχόμενη θητεία. Αυτό μπορώ να σκεφτώ ώστε να επιτύχουμε μια κάποια συνένεση. Γιατί στην περιοχή αυτή με μικρές πλειοψηφίες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα όταν έχουμε τόσο λίγο χρόνο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Κορνίλια για την Ιγκούε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους ε, προηγούμενους ομιλητές και να πω πως ε, χρειάζεται να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και ε, να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην καταπολέμηση και της τρομοκρατίας και στην απομάκρυνση πανάνομου τρομοκρατικού περιεχομένου. Από την άλλη όμως να μην ξεχνάμε την, το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή η ισορροπία νομίζω είναι αναγκαία και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. διότι με την ε, δεδομένη πίεση χρόνου που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Αυτή η εντολή απομάκρυσης, το removal order, είναι ε, αρκετά ασαφές. Πόσο προέκυψε, ποιος αποφασίζει. Θα, χρειάζεται, θα χρειαστεί μια δικαστική εντολή έτσι ώστε να μπορέσει να απομακρυνθεί περιεχόμενο. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη σαφήνεια. διότι παρατηρούμε ότι η διατύπωση παρουσιάζει λήψη σε αρκετά σημεία. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι πρέπει μια δικαστική αρχή ή μια ανεξάρτητη αμερόληπτη αρχή να αποφασίσει για την απομάκρυση του περιεχομένου. Αυτό είναι αρκετά σαφές, το αμερόληπτη ανεξάρτητη αρχή. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη ε, συζήτηση, πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι αυτή η αρχή, τι θα την καθιστά αμερόληπτη και πώς μπορούμε να εγγυηθούμε αυτήν την ουδετερότητα. Μετά, το άρθρο 5, οι αναπομπέ. είναι επίσης ένα προβληματικό σημείο. Θεωρούμε πως ε, το άρθρο αυτό χρειάζεται αρκετή βελτίωση σε ε, σχέση με αυτό που βλέπουμε. Χρειάζεται σαφήνεια σχετικά με την απομάκρυνση περιεχομένου και με την παρούσα διαδικασία δεν βλέπω πώς ε, μπορεί να υλοποιηθεί, διότι χρειάζεται ε, λέει, η πρώτερη συμφωνία με τον ε, επάροχο, με την πλατφόρμα κτλ. Πώς θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τη σωστή συνεργασία. Καλύτερο θα ήταν να διαγραφεί το άρθρο 5, αν συνεχίσει να έχει αυτή τη μορφή στα προδραστικά μέτρα και το άρθρο 6. Εδώ νομίζω πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι τι είναι αυτά τα μέτρα, ποια είναι αυτά. Από τη μία, ναι, θέλουμε ε, να είμαστε προδραστικοί, από την άλλη πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Γι' αυτό χρειάζεται ένα μοντέλο το οποίο θα ακολουθήσουμε σχετικά με τον έλεγχο, ε, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα έπειτα είναι αναγκαίο να γίνει και μία εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με αυτά τα προδραστικά μέτρα. Γι' αυτό με την παρούσα τους μορφή δεν μας ε, ικανοποιούν καθόλου, διότι πιστεύουμε πως δεν συμφωνούν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. νομίζω πως ε, δεν είναι κατάλληλο να προσπαθήσουμε απλά να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Καλύτερα είναι να ε, πάρουμε το χρόνο μας και να εξετάσουμε διεξοδικά το θέμα. Επίσης, ούτε με την οδηγία για την τρομοκρατία, ούτε με κάποια άλλη νομοθεσία μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση ως έχει. Γι' αυτό πιστεύουμε πως δεν είναι κατάλληλη η διατύπωση και ε, της πρότασης αυτής έτσι όπως έχει. Ευχαριστώ πολύ, Κονίλια. Η Εύα Ζολή, ως και οδεσηγήτρια για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δανιέλ Ντάλτον για το σχέδιο γνωμοδότησης, καθώς και τους ε, συναδέλφους για τις προτάσεις τροπολογιών για την απόσυρση αναρτήσεων ε, τρομοκρατικού περιεχομένου. Και εγώ ε, με τις τροπολογίες μου θέλω να ε, προβάλλω την διαφάνεια, την αναλογική δράση και την ασφάλεια δικαίου, ενισχυμένη ασφάλεια δικαίου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει νομική άσκηση. Ε, νομική ασάφεια και δεν θα πρέπει να αποσύρουμε περισσότερες αναρτήσεις από το απόλυτα αναγκαίο. Αυτό αφορά και τις κυρώσεις του κανονισμού, όπως προτείνεται από την Κομισιόν. Θα υπάρχουν αυτοματοποιημένα φίλτρα για το επιγραμμικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε υπερβολικό μπλοκάρισμα περιεχομένου. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την ελευθερία εκφρασής, να υπάρχει αναλογικότητα. Γι' αυτό τα επιπρόσθετα ε, μέτρα των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν το τρομακρατικό περιεχόμενο δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε γενική εποπτεία και φιλτράρισμα. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές που θα επιβάλλουν την ε, απόσυρση θα πρέπει να είναι ε, αυτόνομες ε, και αυτόβουλες και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ειδική νομικού χαρακτήρα μέρημνα. Αν αναγνωριστεί τρομοκρατικό περιεχόμενο θα πρέπει να δοθεί εντολή απόσυρσης. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνει πλήρη σύγχυση. Και εδώ αναφέρομαι στη Europol, η οποία μιλάει για πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι σίγουρα ε, τρομοκρατικές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο αντίστροφο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν έχει θέση σε αυτό τον κανονισμό, γιατί διαφορετικά θα φτάναμε σε μια μεγαλύτερη λογοκρισία στο διαδίκτυο και δεν θα υπήρχε νομική ασφάλεια για τις ε, επιχειρήσεις. Φωνώ με τους προλαλήσαντες ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι σημαίνει τρομοκρατικό περιεχόμενο για να μην γίνει κατάχρηση ως προς την απόσυρση. Υπάρχει η ειδική νομοθεσία κατά πολέμηση τρομοκρατίας που δυστυχώς χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει στη Γαλλία που στρέφεται κατά των πρασίνων που ε, θέλουν να καταπολεμήσουν τα πυρηνικά υπολείμματα και επίσης αυτό αφορά και το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί υπήρξε ένα ειδικό μπλοκάρισμα μεταφοράς ε, χρημάτων μετά από την κρίση του 2008. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς ως προς το περιεχόμενο. Επίσης, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να παρέμβει σε ένα άλλο για να ζητήσει απόσυρση περιεχομένου. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με θέματα κράτους δικαίου, όπως στην Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία. Ελπίζω να μην δεχτούμε εντολές από αυτές τις χώρες για απόσυρση περιεχομένου. Είμαι πεπισμένη ότι έχουμε κοινές ανησυχίες και θα φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό και σε αντίθεση με μερικούς άλλους, θεωρώ ότι θα πρέπει να ψηφιστεί το κείμενο τώρα σε αυτή τη φοιτεία. Θα ήθελα να κάνω και ένα άλλο σχόλιο για την υποκρισία που επικρατεί στην καταπολέμηση της δημοκρατίας και εδώ αναφέρομαι στη δική μου χώρα, τη Γαλλία, η οποία οποία δεν θέλει να εγγραφεί η Σαουδική Αραβία σε χώρες που ξεπλένουν ε, μαύρο χρήμα, καθώς και την απόσυρση των χωρών που είχε, στις οποίες είχε αναφερθεί η Επιτροπή, δηλαδή τέσσερις αμερικανικές χώρες. Μιλάμε για καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω χρηματικών ε, ροών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Ευχαριστώ πολύ, Εύα. Τελευταία ομιλητρία, ένα γκόμες και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλο των σχεδόν εισηγητών. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να συμφωνήσω με το Σεπ Βαζουλή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πώς ε, είναι κάτι το οποίο παραβλέπουμε. Παραβλέπουμε είναι... Δεν είναι αρκετό για να περιγράψουμε αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη. Έχει απόλυτο δίκιο η Birgit Τζίπελ. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ως νομική βάση τον ε, κανονισμό για την ε, ενιαία αγορά. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι πράγματι χρειάζεται μια ανεξάρτητη αρχή, διότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η ελευθερία της έκφρασης και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η... Α, η Νάταλη Γκρισπέκ έχει το λόγο. ε, πολύ σύντομα, καθότι είναι αργά, αλλά είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Αυτό ο φάκελο που επιταχύνθηκε, είναι το ελάχιστο μπορεί να πει κανεί, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και πολύ σημαντικό θέμα. Και για την Επιτροπή μας είναι στρατηγική σημασία προκειμένου να επιχειρήσουμε να ενισχύσουμε τα μέσα μας για την καταπολέμηση της ε, ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο και την προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων και χτυπημάτων μέσω δικτύων που δρούν στο διαδίκτυο. Είναι περίπλοκο ζήτημα και ευαίσθητο. Όλοι οι συνάδελφοι το επανέλαβαν. Εδώ στην Επιτροπή προσπαθούμε διαρκώς να βρούμε την καλή ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως να ανταποκρινόμαστε και τους στόχους της ασφάλειας και στην ανησυχία των ε, συμπολιτών μας. Είναι λοιπόν μια δύσκολη και περίπλοκη ισορροπία, ακόμα περισσότερο ε, καθότι όπως έλεγε και η σκιώδης ομάδος μας η Μάιτε, πρέπει να προχωρήσουμε όπως είπε και η κυρία Ζολή, πρέπει να ψηφίσουμε πριν το τέλος της θητείας. Έχουμε πολλούς τέτοιους φακέλους βέβαια αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ διαρωτούμε ε, μήπως ε, έχουμε ταραχθεί και ε, προσπαθούμε να τρέξουμε εις βάρος της ποιότητας κάποιες φορές. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, εγώ συνάντησα πάρα πολλές ενώσεις ε, ε, νομομαθείς, ε, δικηγόρους, ειδικού για το θέμα αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα στοιχείο το οποίο ίσως δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερα υπό την έννοια αυτή, δηλαδή ο αντίκτυπος για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις και για να είναι σαφής η προσωπική μου θέση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό οι μικρές πύλες, τα μικρά site να συμπεριληφθούν, οι μικρές πλατφόρμες. Αλλά ότι από την άλλη είναι απολύτως απαραίτητο να βρούμε επαρκείς λύσεις. Να παρέχουμε μια συνεχή υποστήριξη, καθοδήγηση σε αυτές τις ε, μικρές επιχειρήσεις Και τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να θεσπιστεί σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος μία αρχή που θα είναι και ανεξάρτητη και αρμόδια γιατί αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει μια διαδικασία πιο ευέλικτη αλλά και πιο σίγουρη σε σχέση με τους στόχους που έχουν τέθει. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα λίγο, νομίζω ότι εντός χρόνου. Ο κύριος Ονίδη νομίζω, λέει ο πρόεδρος, α, η Σοφή, πολύ γρήγορα, αν θέλετε. Κάποια γενικά σχόλια, πρόεδρε, και, να, και σε σχέση και με τα όσα μόλις είπε η Ναταλή, δεν είναι μόνο οι λεπτομέρειες ε, του φακέλου αυτού. Είναι ένας ακόμα από πολλούς φακέλους όπου έχω την εντύπωση ότι μιλούμε για ζητήματα που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ζωή των πολιτών, στις επιχειρήσεις. Και εδώ μιλούμε για την Επιτροπή που ήταν να εστιαστεί όχι μόνο στα μεγάλα και τα σημαντικά. Αν προσθέσετε τα όσα έχουν γίνει τελευταία πέντε χρόνια σε αυτό το πεδίο, σε σχέση με το πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης ή τα μέτρα υπέρ του κλίματος, άλλα μέτρα που έχουμε καθυστερήσει πολύ να αναλάβουμε, όλη αυτή, όλη αυτή η μόδα, η τάση έχει γίνει λίγο ιστερική. Δεν έχουμε αξιολογίες αντικτύπου, δεν έχουμε ακαδημαϊκή έρευνα, δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία από τον ε, επόπτη προστασίας δομένων και τα όσα έχουμε τα αγνοούμε, η Κομισιόν συμπεριφέρεται ως Γενική Γραμματεία των κρατών, των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι 9 στους 10 φακέλους θα απορριφθούν από το δικαστήριο. Και αφήνουμε απλώς όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά στο δικαστήριο. Διότι δεν έχουμε το θάρρος να πούμε, ε λοιπόν, όχι. Φτάνει. Και είναι αλήθεια ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της θητείας που είναι πάντα μια ε, περίοδος, μια στιγμή πίεσης, αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει από το καθήκον να νομοθετούμε σωστά. Σωστά και δίκαια και με πληρότητα. Και μετά από 20 χρόνια ασταμάτητων αντιτρομοκρατικών μέτρων και νομοθετημάτων δεν είχαμε ούτε μία αξιολόγηση, μα ούτε μία, για τα όποια αποτελέσματα εμπετεύθησαν. Είναι απαράδεκτο και είναι και ιδιαίτερα νομικά απαράδεκτο. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα, τα νομοθετήματα θα πρέπει να έχουν, να αποδεικνύουν ότι υπόκεινται στον νόμο της αναλογικότητας. Και ούτε αυτήν την νομική υποχρέωση δεν καλύπτουν. Αφήστε δε την πολιτική. Και εγώ δεν, δεν πραγματικά έχω κουραστεί. Δεν μπορεί να είμαστε όμοιροι αυτής της συνεχούς πίεσης. Θέλουμε να παράσχουμε ασφάλεια στους πολίτες, αλλά όχι και έτσι. Επιταχύνω, Πρόεδρε, γιατί βλέπω ότι αδειμονείται. Ναι, πρέπει να λάβουμε μέτρα ασφαλείας. Έχουμε πάρα πολλές, ε, ε, ε, ε πολλούς ανθρώπους και ομάδες που θέλουν το κακό μας. Όμως πρέπει να ενισχύσουμε και τα πολιτιακά δικαιώματα. Και τα τελευταία 20 χρόνια το μόνο που κάνουμε είναι να υποσκάπτουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Το Εράσμους. Ακόμα και ο ίδιος ο Επίτροπος. Το αποδυναμώνουν. Λιγότερα χρήματα, λιγότερους πόρους, λιγότερη ενίσχυση στους μη καπαόμικρων. Ακόμα και λιγότεροι από αυτού που δίνουμε σε εκείνου που είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να πω πρόεδρε, σκεπτείτε το πραγματικά προτού το ψηφίσετε. Καμία φιλοδοξία. Αυτό βλέπουμε ότι η πρόταση έγινε το Σεπτέμβριο. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο με αυτή τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Ναι, βέβαια χάσαμε χρόνο. Παρότι μετά υπήρξε ταχύτητα. Ε, Πώ θα το έλεγε Μπίργκιτ, δεν θα... Ε, υπήρξε κάποιο, κάποια άλλη μετάφραση, δεν χάσαμε χρόνο. Εκτός μικροφώνου. Δεν χάσαμε χρόνο, πήραμε πολύ χρόνο μέχρι να καταλάβουμε τα πράγματα και τώρα μας πιέζουν να βιαστούμε. Θεωρώ λοιπόν πως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναλογιστεί τι θέλει να πει όταν μας μιλάει για καλύτερη νομοθεσία. Η καλύτερη νομοθεσία πρέπει να είναι αποτελεσματική, να είναι λειτουργική και να σέβεται κάποιους ε, θεμελιώδεις κανόνες. Ναι, βέβαια, η σύγκρουση αρμοδιοτήτων βέβαια δεν είχε να κάνει με το πόσο ποιοτικό ήταν ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, είχε να κάνει με το ε, πόσο ε, δύσκολη μας έκαναν τη ζωή. Αλλά θα δείτε, θα γίνει η ψηφοφορία τέλη Μαρτίου στην Επιτροπή Πολιτισμού και θα δούμε πώς θα πάει. Χάσαμε λοιπόν κάποιο χρόνο και ναι, βια... μας ε, έκανα να βιαστούμε, αλλά όπως και να έχει. Κύριε Ονιντή, θα θέλατε να προσθέσετε κι εσείς κάτι. Δεν ε, είχα προγραμματίσει την σειρά των ομιλητών με αυτή ακριβώς ε, την αλληλουχία ε, έτσι ώστε να σας δώσω το λόγο, αλλά σε πολύ καλό σημείο ήρθε. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω όλους σας, διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό και χρειάζεται να γίνει μια ποιοτική ανταλλαγή απόψεων για την ε, πρόταση. Σήμερα έγινε μια εκδήλωση για τα θύματα τρομοκρατίας. Η Μάιτε ήταν εκεί, θα σας πει αλλά η προστασία των ε, πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με εσάς για την προστασία των πολιτών και μην ξεχνάτε ότι η προσπάθεια πρόληψης περιεχομένου σχετικού με την τρομοκρατία να εμφανίζεται στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική των τρομοκρατών να αναβάζουν τρομοκρατικό υλικό στο διαδίκτυο, τρομοκρατικό περιεχόμενο μάλλον στο διαδίκτυο. Και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών οφείλουν να κάνουν καλύτερη δουλειά, έτσι ώστε να αξιολογείται το περιεχόμενο πιο προσεκτικά. Γι' αυτό και έγινε εκτίμηση αντικτύπου και καταλήξαμε κατόπιν στην πρότασή μας. Νομίζω πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με πολλά από αυτά που είπατε σήμερα και σίγουρα είμαστε γνώμονες για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Βλέπουμε πως ε, αναδύονται κάποια φλέγοντα ζητήματα, πως ε, υπάρχει ανάγκη να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με τον σκοπό της πρότασης αυτής. Οπότε σίγουρα χρειάζεται βελτίωση των ορισμών, όχι μόνο για ε, το περιεχόμενο σχετικό με την τρομοκρατία, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία. Και όπως πρότεινε και η συγκήτρια, χρειάζεται να στοχεύσουμε καλύτερα και όχι περιορισμένα, δηλαδή να μην στοχεύουμε μόνο στην ε, απομάκρυνση του υλικού που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Θα πρέπει ίσως να χρησιμοποιήσουμε και την ε, οδηγία για την καταπολέμηση της δημοκρατίας, την οποία έχετε ήδη εγκρίνει. Έπειτα. Πρέπει να δούμε και το ρόλο των κρατών μελών Γι' αυτό θα θέλαμε να υπάρχει μια κάποια ευελιξία. οι αρχές θα πρέπει να υπόκεινται σε δικαστική εποπτεία, δικαστικό έλεγχο. Αυτό όμως ε, χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και περισσότερη ευελιξία, ε, διότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες ως προς αυτό στα διάφορα κρατημέλη. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια σχετικά με το ποια αρχή είναι η αρμόδια που θα διεξάγει αυτούς τους ελέγχους και χρειάζεται να υπάρχει πλήρης λογοδοσία. Μετά, δεν έχουμε βρει καμία λύση καλύτερη από αυτή που έχετε τώρα ερωπιών σας. Η λύση αυτή είναι σαφής θεωρούμε και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, όμως εξαρτάται και από όλους τους υπολογισμούς της εκτιμής που έχουμε κάνει. Και επίσης σύμφωνα με όλα αυτά, είναι η πλέον κατάλληλη για να αντιμετωπίσει την διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Επίσης, να μην ξεχνάμε τον ε, σημαντικό ρόλο των ε, μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Ε, δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι ούτε και να μην έχουν ευθύνε, όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως χρειάζεται μία κάποια αναλογικότητα ε, ως προς τις κυρώσεις. Τώρα, προδραστικά μέτρα. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι αντίθετα στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και στις αρχές της, ε, για θέματα ευθύνης, θα χρειαστούν διευκρινήσεις με τη μορφή επιστολών, με διάφορους άλλους τρόπους αυτή δεν θα πρέπει να είναι μια υποχρέωση των ε, παρόχων υπηρεσιών, ούτε εκείνη θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ε, συνεχή κατάρτιση και τον έλεγχο, αλλά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πρόσθετες δράσεις έτσι ώστε να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Και Πολλοί από εσά είπατε πως ε, η Ευρωπόλη θα πρέπει να διαδραματίσει πιο ε, σημαντικό ρόλο. Ε, συμφωνούμε απόλυτα. Όχι μόνο η Ευρωπόλη, αλλά γενικά οι, αρχαία, οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία που θα γίνει μέσω διαφόρων διάβλων επικοινωνίας. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει υποχρεωτικός χαρακτήρας. Τόσο ως προς τις υποχρεώσεις και ως προς τις ε, ποινές και τις κυρώσεις. Και ίσως εδώ χρειαστούν περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες και καλύτερη στήριξη προς τις ε, μικρότερες επιχειρήσεις που διαστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη αυτή την πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ονητή. Νομίζω πως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε διότι λείπει και ο κύριος Ντάλτον. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Ευχαριστούμε πολύ και εσά, κύριε Ονίτη. Ελπίζουμε στις 21 Μαρτίου να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που δείχνετε. Έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη πριν ολοκληρώσουμε την ε, συνεδρίασή μας για τις ευρωπαϊκές διαταγές προσκόμισης και δέσμευσης ηλεκτρονικών αποδεκτικών στοιχείων σε ποινικέ υποθέσεις. Η κυρία Ζήπελ έχει συντάξει δύο έγγραφα εργασία με τον Ούνο Μέλο και τους υπόλοιπους κυριώδεις εισηγητές. Ε, μετά Υποβλήθηκαν και άλλα δύο έγγραφα εργασία για τη συνεργασία με, τις, ε, με το δίκαιο τρίτων χωρών. Ε, συντάκτριες ήταν η Birgit Τζίπελ και η Σόφιντ Φέλτ και παρουσιάστηκε και ένα ακόμα έγγραφο εργασία για τι προποθέσει για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΕ από την Birgit Τζίπελ και την Κορνίλια Ένστ. Οπότε ας τα εξετάσουμε. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια για να μας ενημερώσει σχετικά με τη σχέση με το δίκαιο τρίτων χωρών. Μπίργκιτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι αρκετά αργά. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτό το θέμα και ζητώ συγγνώμη γιατί θα χρειαστώ μερικά λεπτά για την παρουσίαση. Θυμόσαστε ότι είχαμε ένα γενικό έγγραφο εργασίας και δύο άλλα νωρίτερα το Φεβρουάριο μαζί με τον Νούνο Μέλο ε, σκιώδη του ΕΛΚ για τη σχέση με τον ε, κανονισμό και τα άλλα ε, κοινοτικά μέσα καθώς ε, και με τους ε, παρόχους υπηρεσιών μαζί με την Κορνίλια Έρνστ. Μαζί με τη Σκιώδη Ιντφελτ και την Κορνίλια Έρνστ από την ΚΟΕ έχουμε συντάξει αυτό το έγγραφο. Γιατί γίνεται αυτή η βάθος ανάλυση του εγγράφου. Σε αντίθεση με το Συμβούλιο που μέσα σε δύο μήνες ε, μίλησε για τη γενική προσέγγιση, το Δεκέμβριο δηλαδή, <coughs> εμείς θεωρήσαμε θα έπρεπε να κάνουμε σε μία εις βάθος ανάλυση της ε, πρότασης και αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα έχουμε συμφωνία πριν από το τέλος της θητείας. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τα ευρήματα από τα τρία έγγραφα εργασίας και με τα δύο επιπρόσθετα είμαι πεπισμένη ότι λάβαμε τη σωστή απόφαση. Ποια είναι τα βασικά ευρήματα το πρώτο έγγραφο μαζί με τη Σόφι Ιντβελ το συντάξαμε σχετίζεται με το κανονιστικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο με τις τρίτες χώρες. Με βάση την ε, ε κοινή αρρωγή Ρωσίας-ΥΠΑ υπάρχει η δυνατότητα πρόσβαση σε αποθηκευμένα στοιχεία στις είπα. σε σχέση με τις ε, συναλλαγές καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Πολύ συχνά αναφέρεται ότι πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι, τεχνικοί και χρηματοδοτικοί. Αυτό αναστρέφει κάπως τη διαδικασία αίτησης δεδομένων με βάση τις ε, δύο τελευταίες ε, κατηγορίες σε σχέση με τους παρόχους και τις εγκληματικές, την έρευνα για εγκληματική δράση υπάρχει συνεργασία μεταξύ παρόχων, ευρωπαϊκών ε, παρόχων και παρόχων από πλευράς ήπα, Άρα ένα νέο μέσον όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ίσως να μην είναι απόλυτα αναγκαίο. Φαίνεται ότι τα προϋπάρχοντα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά εάν τα κράτη-μέλη προσδώσουν τους κατάλληλους ε, πόρους. Επίσης, στο έγγραφο εργασίας λαμβάνουμε υπόψη τη νομοθετική πράξη για τον ΕΦΟΣ, τον ΕΙΠΑ, σε σχέση με μια ενδεχόμενη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης-ΕΙΠΑ. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα σε σχέση με τη νομική βάση για μια τέτοια ενδεχόμενη συμφωνία και πώς μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να συνυπάρξει με τα διάφορα νομικά συστήματα του Cloud Act καθώς και τα, μέσα, τα αποδεικτικά μέσα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ανοιχτά νομικά ε, ζητήματα και δυνάμει του άρθρου 15 ε, και 16 ε, υπάρχει η περίπτωση σύστασης μιας νέας επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και την, ε, τους παρόχους που θα μπορούσαν να βρεθούν σε μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συνεργασία με τρίτες χώρες. Το δεύτερο έγγραφο εργασίας της Κορνίλια Ένστ και μου καλύπτει τους όρους σε σχέση με δύο τέτοια ενδεχόμενα εντάλματα. Εδώ δεν δεχόμαστε την επιχειρηματολογία της Επιτροπής ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο και τις συναλλαγές με βάση τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να προβάλλουν και συγκεκριμένες ε, δράσεις ε, παρακράτησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζητήματα που δεν έχουν τόσο ευαίσθητο περιεχόμενο. Και αυτά μέσα στα πλαίσια της αδειοδότησης. Δεν είναι το ζήτημα ποιος, ότι ποιος μπορεί να προβάλλει ένα ένταλμα, αλλά και ποια θα ήταν τα πλημελήματα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Τα ε, λεγόμενα production orders καθώς και preservation orders μπορούν να ισχύσουν για οποιαδήποτε εγκληματική πράξη. Σε σχέση τώρα με τα στοιχεία συναλλαγής, η Επιτροπή ορίζει ένα κατόφλι λέγοντας ότι ένα τέτοιο αρχικό ένταλμα, production order, αφορά ε, πράξεις ε, οι οποίες α, προέρχονται από κράτη όπου υπάρχει κράτηση που ισχύει για τουλάχιστον τρία χρόνια. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει μια δυτή αρχή εγκληματικότητας και φαίνεται ότι αυτό το κατόφλι οδηγεί στην κατάρρευση των πάντων. Με βάση τα προηγούμενα έγγραφα λοιπόν φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό ε, το μέσον άμεσης εφαρμογής κυρωτικού πλαισίου βρίσκεται πέρα από τα ευκταία δεδομένα. Αυτό αφορά και την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, αυτό ε, εκτιμάται μόνο από την αρχή αδειοδότησης. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, υποχρεωτικής κοινοποίησης μεταξύ της αρχής ε, κοινοποίησης και των κρατών μελών όπου υπάρχουν υπάροχοι. Έτσι το κράτος εκτέλεσης θα ε, μπορέσει να εκτελέσει τις πράξεις μόνο όταν δεν υπάρχει η δυτή αρχή ε, σε σχέση με εγκληματικές πράξεις. Υπάρχουν και άλλα δύο έγγραφα εργασίας, τα οποία τώρα επεξεργαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια εις βάθος ανάλυση της πρότασης. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την επιφανειακή εξέταση όπως έκανε το Συμβούλιο και όπως μας επέβαλε η Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Μπίργκιτ. Η, η Σόφη. ναι, Πρόεδρε. Κάποια πρόσθετα σύντομα σχόλια. Ο κατάλογος των νομικών ζητημάτων και ερωτηματικών είναι μακρύς και το καθιστά σαφής ότι η πρόταση αυτή δεν είναι όριμη. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί. Να πω αμέσως για να είμαι σαφής, ότι είμαι υπέρ της αρχής της δημιουργίας αυτής της κοινή περιοχής νομικής και αστυνομικής συνεργασίας. Καθότι φεντεραλίστρια είμαι. Αλλά πρέπει να έχουμε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις και αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Δεν ξέρω δηλαδή από πού να αρχίσω. Ποιος αποφασίζει είναι σχεδόν αντισυνταγματικό για να το πω έτσι να το αφήνει κανείς σε μια επιχείρηση να αποφασίζει κατά πόσο είναι έτοιμα είναι δικαιολογημένο ή όχι. Οι πάροχοι λένε εμείς δεν μπορούμε καν να αποφασίσουμε διότι δεν ξέρουμε ποια είναι η δικαιολόγηση του αιτήματο. Αυτές τις πληροφορίες δεν τις λαμβάνουμε και επομένω πώς θα κρίνουν οι πάροχοι. Και αν έχοντας κάνει μία πλήρη ανάλυση που την πλήρη ανάλυση την περιμένουμε μήνες από την Κομισιόν, αν τους χρειαστεί εβδομάδες, πάλι αδύνατον θα είναι. Αφήστε δε που δεν θα έπρεπε να αποφασίζουν αυτοί, να εξαρτάται από αυτούς. Και δεν είναι τρόπος αυτός να αντιπαραθέτει κανείς ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα έναντι ε, των συμφερόντων των κρατών μελών. Επίσης ως προς τα αποδεκτικά στοιχεία εργαζόμαστε υπό την υπόθεση ότι τα δικαστικά συστήματα, τα συστήματα δικαιοσύνης κρατών μελών είναι ισότιμα. Αλλά υπάρχει κράτος μέλος που έχει ξεκινήσει διαδικασία άρθρο 7, όπως και το Κοινοβούλιο, διότι θεωρούμε ότι οι δικαστικές αρχές δεν είναι ανεξάρτητες, τότε τι θα γίνει. Μια χώρα που λαμβάνει αίτημα από την Πολωνία τι πρέπει να πει λυπούμεθα αλλά αρνούμαστε το έτοιμά σα. Και αν δείτε τις αποφάσεις του δικαστηρίου, ούτε καν οι δικαστές δεν μπορούν να αρνηθούν ένα, για παράδειγμα, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Περιμένουμε ότι θα αρνηθούν λοιπόν οι επιχειρήσεις. Είναι τελείως παράλογο αυτό. Οι προθεσμίες είναι πολύ στενές, οι εγγυήσει είναι ανεπαρκείς, η διατλαντική διάσταση είναι απολύτως προβληματική. Δηλαδή το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί την πρόταση αυτή στο τραπέζι, ήταν σαφής ακόμα και πριν το κάνει αυτό, ότι ο τελικός στόχος ήταν η Διατλαντική Συμφωνία. Ώστε να έχουμε μια νομική βάση, ένα πλαίσιο για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε από την αρχή αλλά νομίζω κοροϊδευόμαστε. Ως προς την διατλαντική διάσταση πρέπει να επενδύσουμε σημαντική προσπάθεια για να βελτιώσουμε το παρόν πλαίσιο συνεργασίας και μέχρι να έχουμε εξαντλήσει τα έμλατς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διατλαντικές συμφωνίες σε αυτό το επίπεδο. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Για την δε εσωτερική διάσταση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνώ πολύ με την αρχή, αλλά προηγουμένως πρέπει να έχουμε τι εγγύσει. Και μετά πρέπει να έχουμε και μια πληρέστατη υδατοστεγανή πρόταση για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και αυτή εδώ οπωσδήποτε δεν καλύπτει τέτοιες προϋποθέσεις. Πρόεδρος, ήθελα να, απλώς να σας πω ότι πολλά από τα σημεία αυτά τα αναφέραμε με το Συμβούλιο ε, στις επαφές για τα έμλατς, για το τι πρέπει να κάνουμε με αυτά προτού προχωρήσουμε, αλλά ε, φαντάζεστε ότι κάποια κράτη-μέλη του Συμβουλίου είναι πραγματικά σημαντικά ως προς αυτό. Εγώ κατέστησα τη θέση πάντως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαφή, η Κορνίλια. Μάλιστα. Έχουμε και ένα άλλο δημιούργημα, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όπως είπαν και οι συνάδελφες, νομίζω, συνάδελφοι, νομίζω πως χρειάζεται βελτίωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι αποδεκτό. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι το χάος ε, αποτελείται από την πληθώρα κατηγοριών που υπάρχουν, ε, τα στοιχεία που δεν είναι σωστά ταξινομημένα, ε, τις διάφορες εντολές για την εκτέλεση των οποίων κανείς δεν ξέρει ποιος είναι αρμόδιος. Εδώ μπλέκονται πολλά. Από τη μία οι κατηγορίες των δεδομένων, από την άλλη οι αρμοδιότητες για την διατήρηση των στοιχείων ή για την ε, υποβολή των στοιχείων αυτών. Και μην ξεχνάτε πως ε, υπάρχουν 27, σύντομα 27 διαφορετικά κράτη-μέλη με διαφορετικές διαδικασίες το καθένα. Θα μπορούσαμε λοιπόν, γενικεύοντας ε, τα πράγματα αρκετά, να πούμε ότι αυτός αυτή η πρόταση δεν θα βελτιώσει την κατάσταση, μάλλον θα την επιδεινώσει. Ας δούμε τι γίνεται με τα δικήματα. Ήδη έχει ακουστεί ότι η έννοια του αδικήματος ενδιαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και αν δούμε την ε, κατάσταση πιο προσεκτικά θα δούμε ότι το διπλό αδίκημα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, όχι μόνο από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αλλά και πολλές φορές ε, μέσα σε ένα ίδιο κράτος μέλος. Στη Βαυαρία, ας πούμε, διαφορετικά από ότι στην ε, υπόλοιπη Γερμανία. Αυτά σε ό,τι αφορά το διπλό αξιόπινο. Ε, μετά υπάρχουν και άλλα θέματα περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης, και πρέπει να δούμε ότι εάν θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στο διπλό αξιόπινο, τότε θα παραμελήσουμε και ίσως ε, θα ε, συρρυκνώσουμε ορισμένα άλλα δικαιώματα. Ας δούμε τώρα με περισσότερη προσοχή την ε, πρόταση και ας τη συγκρίνουμε με τις άλλες εντολές. Ας δούμε τι γίνεται με την αναλογικότητα. Ε, με τους ε, κατηγορούμενους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στους ε, άλλους κανονισμούς, στο ότι υπάρχει κάποια σχέση αιτίου και αιτιατού. Εδώ πέρα δεν βλέπουμε καμία σχέση. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες ελεύθερες έτσι, διατυπώσεις αυθαίρετες που δεν στηρίζονται πουθενά. Επίσης, το δικαίωμα προσφυγής ε, δεν αναφέρεται στην πρόταση. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην ε, δικονομία, στην δικονομική διαδικασία, το τι μπορεί να κάνει κάποιος σε ποια περίπτωση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες λοιπόν ως προς τη διαδικασία. Γι' αυτό ας αναρωτηθούμε εάν αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας είναι ένα κείμενο που πρέπει να δεχτούμε ή απλά να τα απορρίψουμε. Χρειάζεται ένα δεσμευτικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ κρατών μελών, έτσι ώστε να αναγκαστούν να συνεργαστούν με σαφείς κανόνες. Ε, θα πρέπει επίσης να υπάρχει το δικαίωμα ε, της άρνησης εκτέλεσης μιας εντολής κατόπιν αιτιολόγησης και θα πρέπει σε όλα αυτά να υπάρχει αναλογικότητα. Ε, υπάρχουν λοιπόν τόσα πολλά προβλήματα και τόσες πολλές ελλείψεις που νομίζω πως μπορούμε να το συζητάμε αυτό για πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και την ε, Κονίλια, την ε, Σοφίν Φέλτ και την Πίργκιτ Τσίπελ για την παρουσίαση. Θα ήθελε κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Θα παρουσιάσουμε τώρα στις 2 Απριλίου τα υπόλοιπα δύο έγγραφα εργασίας και αν το θελήσει η κυρία Μέη θα είμαι και εγώ εδώ για να, το, για να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Αλλιώς λυπάμαι πολύ αλλά δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Κορνίλια θα μου λείψεις. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τους πρωθυπουργούς. Α, ναι, 18 Μαρτίου, επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σίγουρα θα είμαι εδώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το βασιλείο της Ισπανίας, αλλά μάλλον δεν θα έπρεπε να αναφερθώ σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ τους εδερμηνείς και το υπόλοιπο προσωπικό. Θα τα πούμε αύριο.